Good afternoon, colleagues, and I'm sorry for the short delay. We have a quite a short meeting. Καλησπέρα, συνάδελφοι. Έχουμε μικρή ε, μέρη διάταξη. Τρία θέματα πολύ ενδιαφέροντα βέβαια. Πρώτον, θα ήθελα να ευχαριστήσω, να καλωσορίσουμε την ε, Λούισα Μπέρς από την υπηρεσία του ΟΗΕ για τη μετανάστευση η οποία και θα μας παρουσιάσει την τρέχουσα κατάσταση για την, το, δημόσιο, το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ε, τυπική και μετανάσταση. μετανάστευση. Επίσης έχουμε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης κυρία Νούτσεν η οποία, την οποία την είχαμε και πρόσφατα εδώ μαζί μας και είναι και ο κύριος, μαζί μας είναι ο κύριος Αμπρόζη από τον Διεθνή Οργανισμό για τη μετανάστευση Στην Ολομέλεια του ΟΗΕ της 19 Σεπτεμβρίου ε, παρευρέθησαν πολλοί ευρωβουλευτές όπου και συζητήθηκε το ζήτημα των μεταναστών και των προσφύγων και αποφασίστηκε να δοθεί καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις. Και ο τίτλος του εγγράφου που προέκυψε ε, είναι η διακήρυξη της ε, Νέας Υόρκης. Ήταν μεγάλη η αντιπροσωπεία, η κυρία Βίκστρομ, η κυρία Εγγράφεν και η κυρία Έλλη Σλάιν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μπορούσα να πω πολλά ακόμη για το σύμφωνο αυτό Καλύτερο όμως να ακούσουμε την Λουίς ε, Άρμπουρ που θα μας ενημερώσει χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για θέματα μετανάστευσης. Κύριε Άρμπουρ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ για να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση για τη διαδικασία ανάπτυξης του Παγκόσμιου Συμφώνου για την Μετανάσταση. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ατομικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους άλλους ομιλητές που βρίσκονται εδώ σήμερα για αυτό που ελπίζω ότι θα είναι μια ειλικρινής και γόνιμη συζήτηση. Η μετανάσταση είναι η ιστορία της ανθρωπότητα από τις απαρχέ της ε, είναι η ιστορία ορισμένων εξημών εδώ στην αίθουσα, είναι η ιστορία ε, γυναικών, ανδρών, παιδιών που έχουν ζητήσει, αναζητήσει νέους ορίζοντες, ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Η εμπειρία αυτή είναι οικία σε πολλούς ε, Ευρωπαίους. θα ήθελα γι' αυτό να σας ακούσω και να συμμετάσχω σε έναν επικοδομητικό διάλογο. Θα ήθελα παρόλα αυτά να αναγνωρίσω τις πραγματικές προκλήσεις που το ζήτημα της μετανάστευσης ε, συνιστά ε, για χώρες και τοπικές κοινωνίες ολόκληρο τον κόσμο. Οι κινήσεις ανθρώπων που παρατηρούμε σε όλο τον κόσμο, στην Κεντρική Αμερική, στην Νοτιοανατολική Ασία, την Αφρική, έχουν προκαλέσει ε, σημαντικές ανησυχίες. Είναι σαφές ότι η απουσία επί της αρχής και συνεργατικής μετανάστευσης και της διακυβέρνηση αυτής σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο ευθύνεται για την τρέχουσα κατάσταση. Αυτό που αντιμετωπίζουμε δεν είναι ακριβώς μεταναστευτική κρίση, αλλά μια κρίση ως προς τη διαχείριση της μετανάστευσης και είναι προφανώς και μια κρίση αλληλεγγύη. Αυτό λοιπόν έφερε τους αρχηγούς ε, ε, κρατών και κυβερνήσεων ε, στην ε, Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πέρυσι το Σεπτέμβριο για να συζητήσουν πώς η διεθνής κοινότητα μπορεί να απαντήσει σε αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο της μαζικής μετακινήσεων προσφύγων και μεταναστών. Στην ε, εμβληματική λοιπόν διακήρυξη της Νέας Υόρκης, Νέας για, πρόσφυγες, για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες αναγνωρίζουν ότι απαιτείται επιτακτικά καλύτερη παγκόσμια συνεργασία στη διακυβέρνηση της μετανάστευσης. Πρόκειται για ένα ιστορικό έγγραφο ε, δέσμευσης πολιτικής προκειμένου να εξασφαλιστεί ε, η ασφαλής, ομαλή και τυπική μετανάστευση με ε, σεβασμό στις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με επίκεντρο τον άνθρωπο, με βάση στοιχεία πραγματικά και όχι με βάση τις επιθυμίες διαφορών πλευρών. Η ε, η διακυβερνητική διάσκεση η οποία ξεκίνησε με αυτή τη διακήρυξη Νέας Υόρκης ε, και η οποία θα ολοκληρωθεί το, στα τέλη του 2018 θα καταλήξει στην έγκριση του Παγκόσμιου Συμφώνου για την ασφαλή, ομαλή και τυπική μετανάστευση. Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων συμμετείχαν ε, ε, πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς, κοινωνία των πολιτών, φυσικά οι κυβερνήσεις, ε, εργατικά κινήματα και άλλοι. Να σας πω λοιπόν κάποιε παρατηρήσεις σχετικά με τι διαβουλεύσει που βρίσκονται σε εξέλιξη μέχρι στιγμής. Αυτές θα επικεντρωθούν στα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των μεταναστών, την αντιμετώπιση της ξενοφοβίας, την αντιμετώπιση των ριζικών αιτίων της μετανάστευση, καθώς και το ζήτημα της διεθνού συνεργασία και διακυβέρνηση ε, του φαινομένου τη μετανάστευση στραφώ στο πρώτο θέμα, ανθρώπινα δικαιώματα όλων των μεταναστών. Το διεθνές νομικό πλαίσιο ήδη προβλέπει ε, τις βάσεις πάνω στην οποία θα βασιστεί αυτό το παγκόσμιο σύμφωνο. Τα κράτη-μέλη επανεπιβεβαίωσαν στην διακήρυξη της Νέα της ότι όλοι οι μετανάστες, ανεξάρτητα από το καθεστώς υπό το οποίο βρίσκονται, έχουν δικαιώματα. Παρά το γεγονός όμως ότι υπάρχει στιβαρό διεθνές δίκαιο και υπάρχει και η δέσμευση πολιτική να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της μετανάστευσης με επίκεντρο τον άνθρωπο, υπάρχει ένα κενό ως προς την εφαρμογή. Και ιδίω ε, αυτό το κενό αφορά την προστασία των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στέγαση, εκπαίδευση, δικαιοσύνη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η παράτυπη μετανάστευση ε, ενισχύει την ε, ευαλωτότητα των μεταναστών σε με πάρα πολλούς τρόπους. Με δυσανάλογο τρόπο ε, είναι εκτεθειμένοι οι μετανάστες σε διακρίσεις, περιθωριοποίηση και κακομεταχείριση. Πολλοί εργάζονται κάτω από συνθήκες εκμετάλλευσης, ε, φοβούμενοι τον, τον κίνδυνο της απέλασης. Είναι πολύ πιθανό ε, πολλοί άνθρωποι από αυτούς φοβούνται να καταγγέλουν εγκλήματα που διαπράττονται εναντίον τους. Το να δημιουργηθούν τύχοι ε, ανάμεσα στην ε, επιβολή των, το, το, της νομοθεσίας για τη μετανάστευση και, και, τους, και τις δημόσιες υπηρεσίες είναι ένας ε, αποτελεσματικός τρόπος για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην, ε, στην, ε, στο δικαίωμα άσκησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ αυτών η δικαιοσύνη, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εκπαίδευση. Κάποιοι από τους μετανάστες πολλές φορές αντιμετωπίζουν ένα καθεστώς πολύ ψηλής ευαλωτότητας. Δεν είναι απλώς οικονομικοί μετανάστες. Αυτή η απλουστευτική προσέγγιση δεν ε, ανταποκρίνεται ούτε στην περιπλοκότητα των λόγων που ε, οδηγούν ανθρώπους να μετακινούνται, ούτε και στην προστασία που χρειάζονται. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για ε, γυναίκες και κορίτσια που αντιμετωπίζουν κινδύνους, ασυνόδευτους, ασυνόδευτα παιδιά, ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες. Πρέπει να επανεπιβεβαιώσουμε και στην πολιτική και στην πράξη την θεμελιώδη σημασία του σεβασμού, της προστασίας και της ικανοποίησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των μεταναστών ανεξάρτητα από το καθεστώς τους. Όσον αφορά τώρα ε, την αντιμετώπιση ε, της ξενοφοβίας. Παρά την, ε, τα δηλητηριώδη σχόλια που ακούγονται, η μετανάστευση δεν πρέπει να θεωρείται ως πρόβλημα που πρέπει να επιληθεί. Η μετανάστευση μπορεί να είναι μια εμπειρία για πολλούς ανθρώπους που τους ενδυναμώνει. Μπορεί επίσης να συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση κάποιων από, το, κάποιων από τις πιο δύσκολες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας. Η κλιματική αλλαγή, βιώσιμη ανάπτυξη, μείωση πληθυσμού, γύρανση του πληθυσμού. Η μετανάστευση έχει αναγνωριστεί ως μια ε, προδραστική στρατηγική προσαρμογής, ε, μια, ε, ένα φαινόμενο που μπορεί να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και ως όχημα για την ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα των φίλων. Είναι σημαντικό να αμφισβητήσουμε κάποιες από τις κυρίαρχες αντιλήψεις όσον αφορά τη μετανάστευση, μύθους αλλά και εσφαλεμένες αντιλήψεις που πολλές φορές αναπαράγονται καθημερινά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ωστόσο, οι αυξημένες προσπάθειες για τη συλλογή και την κοινοποίηση των σχετικών δεδομένων είναι μόνο ένα μέρος αυτής της εξίσωσης. Πρέπει οι προσπάθειες αυτές να ε, αντιστοιχιστούν με την επιθυμία να αναγνωριστούν οι, οι πραγματικές ανησυχίες που, ε, στις οποίες βασίζονται οι αρνητικέ αντιδράσεις στην μετανάστευση. Οι απαντήσεις που, μπορούν που θα δοθούν δεν μπορούν να είναι απλουστευτικές. Αν δεν καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες αυτές, ο, διά, ο διάλογός μας θα είναι διχαστικός και δεν θα φέρει αποτελέσματα. Δεν θα αυξήσει τη δημόσια υποστήριξη για τις αντίστοιχες πολιτικές που απαιτούνται. Αντιθέτως, μπορεί τα πράγματα να πάρουν και πολύ άσχημη τροπή. Γι' αυτό και θα ήθελα να καλέσω τους ευρωβουλευτές σήμερα να ηγηθούν των προσπαθειών για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και της ξενοφοβίας ε, προκειμένου να μπορέσει να γίνει ένας ισορροπημένος και χωρίς διακρίσεις διάλογος που θα βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία που θα αντιμετωπίζει και θα απαντά στις ανάγκες τόσο των μεταναστών αλλά όσο και των ε, κοινοτήτων, κοινωνιών που τους φιλοξενούν. Ποια είναι τα ριζικά αίτια της μετανάστευσης. Παρατηρούμε καθημερινά την απελπισία πολλών γυναικών, ανδρών και παιδιών που αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολες και αντίξωες συνθήκες, τραυματισμούς, ακόμα και τον θάνατο, καθώς αναζητούν μια καλύτερη ζωή. Τα κίνητρα για να κάνει κανείς τέτοια ταξίδια είναι πολύ περίπλοκα. Πολλοί άνθρωποι ε, φεύγουν ε, βάσει πραγματικά της δικής τους επιθυμίας, άλλοι όμως αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους για να, για να ξεφύγουν από τον πόλεμο, τις διώξεις, τις διακρίσεις, την ε, επισφάλεια όσον αφορά την, ε, την, ε, την τροφή, τη φτώχεια και την κλιματική αλλαγή αλλά και άλλους λόγους. Σε πολλές, φορές, σε περιπτώσεις μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι εθελοντικά φεύγουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες από τις αιστείες τους. Ωστόσο, η γραμμή που χωρίζει εκείνους που φεύγουν εθελοντικά και εκείνοι που αναγκάζονται να ε, εγκαταλείψουν τις τους είναι θολή. Γεγονός είναι πάντως ότι όλοι οι μετανάστες πρέπει να απολαμβάνουν των δικαιωμάτων τους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την, τις ανάγκες προστασίας που, των μεταναστών χρειάζεται να, κατανοήσουμε και να αξιολογήσουμε για ποιο λόγο μετακινούνται οι άνθρωποι. Η διεθνή κοινότητα πρέπει να ε, επιταχύνει την, ε, τις δράσεις της προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ριζικά αίτια της, της μετανάστευσης. Όταν όλοι οι παράγοντες που οδηγούν στη μετανάστευση, για παράδειγμα ε, η μεγάλη και άτυπη ανεπίσημη αγορά εργασίας που ενθαρρύνει τις μετακινήσεις, όταν όλοι οι παράγοντες αντιμετωπιστούν, ε, ε, θα, θα, θα αποδειχθεί ότι το να σηκώσουμε κι άλλα εμπόδια στην πραγματικότητα το μόνο που κάνει είναι να αυξάνει τον κίνδυνο για τους ανθρώπους που μετακινούνται. Διεθνή συνεργασία και διακυβέρνηση. Είναι κρίσιμο σημείο να υπάρξει διεθνής συνεργασία και διακυβέρνηση του φαινομένου της μετανάστευσης ε, μόλις ε, ε, τεθεί σε ισχύ αυτό το παγκόσμιο σύμφωνο. Θα πρέπει η συνεργασία να οδηγήσει στην ικανότητα των κρατών να, διακυβέρ, να, διαχειρίζονται τα σύνορά τους. Οι προσπάθειες για την, για τον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης ε, μέσω των συνεργειακών ελέγχων των απελάσεων και των επιστροφών όχι μόνο έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές ε, ως μορφές αντιμετώπισης αλλά έχουν ε, δυσκολεύσει πολλές φορές σε πολλές περιπτώσεις την ανάπτυξη μιας, ε, ενός πνεύματος αλληλεγγύης τόσο από την πλευρά των κυβερνήσεων όσο και από την πλευρά των κοινωνιών μέτρα όπως ε, η ποινικοποίηση της ε, παροχής βοήθειας και της ανθρωπιστικής ε, συνδρομής σε, παράτιμους, σε μετανάστες μπορεί να έχει ε, ακούσιες αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο για τους ίδιους μετανάστες αλλά και για όσους καλή την πίστη προσπαθούν να προσφέρουν αυτού του είδους τη βοήθεια. Πολλές φορές η βοήθεια αυτή προσφέρεται αναγκαστικά χωρίς τις απαραίτητες εγγυήσει και καταλήγει και σε ποινικά μέτρα εναντίον αυτών που τη δίνουν. Το να εξασφαλιστούν και να εξευρεθούν ε, εναλλακτικέ ε, προς την ε, κράτηση και ιδίως των παιδιών είναι μία από τις δεσμεύσει που ανέλαβαν τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ στην διακήρυξη της Νέα Υόρκη. Μέσω της διευκόλυνση ασφαλέστερων εναλλακτικών στα επικίνδυνα ταξίδια και εξασφαλίζοντας ε, εργατική κινητικότητα, εκπαίδευση, επανένωση οικογενειών, μπορούμε να ε, μειώσουμε την ανάγκη άνθρωποι να κάνουν ε, το ταξίδι της μετανάστευσής τους μέσα από παράτυπες οδούς. Με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί και το, η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ικανότητα των, των ε, κυβερνήσεων να διαχειριστούν το ζήτημα, το φαινόμενο της μετανάστευσης. Είναι ε, πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι ε, η νομοθεσία ευρωπαϊκή βασίζεται στις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Ξέρω ότι είμαστε μαζί σε αυτόν τον αγώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, πρόσκληση που μου απευθύνατε και προσβλέπω σε μια γόνιμη και επικοδομητική συζήτηση σήμερα. Θα ήθελα να κάνετε πιο αυθόρμητες, ε, αυθόρμητα μάλλον χειροκροτήματα. Ας είσαστε λίγο πιο ανθρώπινοι, ήταν, θα ήταν μια καλή ευκαιρία να δείξετε τώρα ανθρωπιά. Ευχαριστούμε, δικαστή Άρμπορ. Θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις για την εμπειρία σας. Και υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι που είναι εδώ. Κάτι θέλω να πω για την προσέλευση. Είναι απόγευμα, είναι 3.30 το, το απόγευμα. Συχνά χαλαρώνει η προσέλευση. Ε, σας ευχαριστούμε για αυτά που είπατε και χαίρομαι που είναι εδώ ε, που είναι εδώ η συνάδελφος από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, που είναι ε, η Διευθύντρια για το Human Rights Global. Η Λότη θα πάρει το λόγο για περίπου 7 λεπτά. Συμφωνεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για το Παγκόσμιο Σύμφωνο. Από την, μετά την πολύ επιτυχή συνεισφορά σας ε, πέρυσι στη Σύνοδο Κορυφής, είναι σημαντικό να παραμένετε δραστήριοι μέσω, μέσω, μέσω διαφορών ενημερώσεων. Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί με τη Λουίζα Άρμπορ στο Δήμα. Είναι ένα πρόσωπο κλειδί ως εκπρόσωπος ε, του Γενικού Γραμματέα για τη Μετανάστευση και στη διακυβερνητική διάσκεψη θα συμμετάσχει και θα εκπροσωπήσει τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Επίσης, ο κύριος Σαμπρόζιο. Ε, συνεργαζόμαστε στενά σε μια δέσμη θεμάτων με τον κύριο Αμπρόζη Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη χθεσινή διάσκεψη, για την διάσκεψη. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ε, στα πλαίσια του, της Συνόδου Κορυφής, μιλάνε για την μετανάστευση. Όπως είπε η Λουίζα Άρμπορ, είναι μια πραγματικότητα η μετανάστευση, δεν θα τα ξαναπώ όλα αυτά. Ε, είναι σωστό να μην τη λέμε κρίση. Να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο κρίση και να εξετάσουμε καλύτερα πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τη μετανάστευση με έφτακτο, ασφαλή και σίγουρο τρόπο, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη προστασία και τα δικαιώματα. Η ανθρώπινη κινητικότητα υπήρχε απαρχαιωτά των χρόνων. Και νομίζω ότι το G20 ε, δημιούργησε μια ομάδα εργασίας για την ανθρώπινη κινητικότητα, γιατί ε, προσπαθ το να το καταστήσουμε ένα διεθνές θέμα και να μην θεωρηθεί ως ένα πρόβλημα αποκλειστικά της Ευρώπης και της Αφρικής και να θεωρηθεί παγκόσμιο θέμα που μας αφορά όλους με παγκόσμια ε, επιμερισμένη ευθύνη στην Ασία, στην Νότιο Αμερική κτλ. είναι πολύ σημαντικό. Ε, είμαστε σε έναν κόσμο με 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ε, το να μετακινούμαστε και να περνάμε τα σύνορα είναι ανθρώπινη φιλοδοξία. Πρέπει να έχουμε κάποια διακυβέρνηση της ε, μετανάστευσης. Και νομίζω μόνο σε παγκόσμιο επίπεδο θα, βάλουμε, θα προωθήσουμε τα μέτρα παγκόσμιας διακυβέρνησης. Ε, φυσικά υπάρχουν εκατοντάδες τρόποι για να το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε πολλά να μάθουμε από την Αφρική, από την Ασία, όπου οι χώρες έχουν ε, συγκεντρώσει διαφορετικές ε, εμπειρίες και διδάγματα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό στα πλαίσια του Παγκοσμίου Συμφώνου να μοιραστούμε όλες αυτές τις εμπειρίες. Φυσικά η μετανάστευση δεν πρόκειται να φύγει ε, λόγω της αστάθειας των χωρών κτλ. κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε το σύμφωνο αυτό για τη μετανάστευση ως μια ευκαιρία για να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα κινητικότητας για τους ανθρώπους, μια και να το παρουσιάσουμε με μια θετική χρειά, ως θετικό αφήγημα. Το χρειαζόμαστε αυτό. Να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη κλίμακας μετακινήσεις. Ε, νομίζω ότι η εξωτερική πτυχή της ε, μετανάστευσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την ε, διαχειριζόμαστε και μαθαίνουμε πάρα πολλά από τις εταιρικέ σχέσεις και τις συνεργασίες που έχουμε, ε, που ελπίζουμε αυτή την εμπειρία τη μεταφέρουμε και στον ΟΗΕ. Είναι όντως μια διακυβερνητική διάσκεψη. Ε, Μεξικανοί και Σουηδοί ε, επικεφαλής ε, διαχειρίζονται τη συζήτηση αυτή στο επίπεδο του συμφώνου. Εγώ θα έλεγα να μην υπάρξουν νέες δομές, θα ήθελα να γίνουμε πιο φιλόδοξοι επί της ουσίας και φυσικά θα πρέπει να δοθεί και κάποια συνέχεια, ένα follow-up ε, που θα συνοδεύει τη δράση, ούτω ώστε να μην γίνει μια εκδήλωση ξεκομμένη. Ε, το να μιλήσουμε για ευκαιρίες που μας περιμένουν ε, σημαίνει ότι είναι τμήμα μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής ε, θεώρησης ε, με διαφορετικά μέτρα σε διαφορετικές φάσεις της διαδικασίας ε, μαζί με, όπως και οι SDGs, οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, ε, ε, τα επόμενα 15 και 20 χρόνια θα μας συνοδεύει και θα μας καθοδηγεί σαν πηξίδα σε αυτά που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Η περσινή δήλωση ε, της Νέας Υόρκης ήταν πάρα πολύ φιλόδοξη, ήταν πολύ καλή, παρότι θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες μας με πιο καλό τρόπο. Επίσης θα πρέπει να κάποια στοιχεία της δήλωσης της Νέας Υόρκης να τα κάνουμε λίγο πιο επιχειρησιακά και πιο στοχοθετημένα. Επίσης, λοιπόν, θα πρέπει να τονίσουμε όλες τις ευκαιρίες, αλλά και βεβαίως τις προκλήσεις. Είναι ακόμα η αρχή της διαδικασίας. Θα πρέπει να έχουμε ένα ισορροπημένο κείμενο. Τελικά, είναι σημαντικό να θεωρούμε ότι είναι δικό μας κείμενο. Εμπλέκονται 193 χώρες, όλες θα πρέπει να εμπλακούν πραγματικά και χρειαζόμαστε ένα κείμενο που τελικά θα είναι θετικό για όλους. Και θα υπάρξουν βεβαίως κάποια δούνε και λαβήν, ε, κάποιοι συμβασμοί, αλλά κάτι θετικό για όλους θα πρέπει να υπάρχει. Θα πρέπει να βρούμε κοινό έδαφος, ε, να γίνουν συγκλήσεις. Είναι μια διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει. ούτως ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα τελικό που θα έχει κάτι θετικό για όλους. Γιατί μην ξεχνάτε ότι και η προθεσμία είναι πάρα πολύ σφιχτή. Όπως είπε η κυρία Αν θέλουμε να πετύχουμε συμφωνία του χρόνου, πρέπει να κάνουμε πολλά τώρα. Ε, πρέπει να μάθουμε πολλά από τις εταιρικέ σχέσεις πλαίσια. Ε, εμείς στη σχέση μας με τις τρίτες χώρες έχουμε πολλές εταιρικές σχέσεις. Υπάρχει αυτή η ιδέα των εταιρικών σχέσεων ότι πρέπει να βρούμε τρόπους για να οργανώσουμε τις σχέσεις που να έχουν στοιχεία θετικά και για τους ε, δύο εταίρους. Στα πλαίσια μια σχέση πάντα. Δεύτερον, θα πρέπει να κινηθούμε συνεντικά. Αυτό σημαίνει εν μέρη να βασιστούμε σε αυτά που έχουμε τη δήλωση της Νέας Υόρκης, το αποτέλεσμα της θεματικής διαβούλευσης, που είναι τώρα στον τρίτο γύρο και που λειτουργεί απόλυτα ικανοποιητικά, με έντονη παρουσία των κρατών, και πάρα πολλές όμως ε, ΜΚΟ και οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών που εμπλουτίζουν τη συμμετοχή. Θα πρέπει επίσης με τις χώρες εταίρους να εξασφαλίσουμε ότι όλοι βάζουμε κάτι στο τραπέζι. Γιατί αν κοιτάξουμε τις χώρες του κόλπου, οποιαδήποτε περιοχή, τις ασιατικές χώρες ή τις χώρες ΑΖΕΑΝ, όλοι έχουν εμπειρίες, έχουν κάποιες πρακτικές, κάποια μαθήματα, διδάγματα που μπορούν να μας εμπνεύσουν. Και νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Νομίζω ότι η περιφερειακή διάσταση λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να τροφοδοτήσει τη διαδικασία. Τρίτον, θα πρέπει να μιλήσουμε με πολλούς εταίρους, όπως και στον ΟΗΕ. Ε, και εμείς έχουμε μία, έχουμε μία σειρά από διαλόγους, κανάλια, εργαλεία, έχουμε παγκόσμιες σχέσεις. Μπορούμε να κάνουμε την, προσ... την έξτρα προσπάθεια να πάμε προς, αυτές, προς, το... προς την μεριά εκείνων των χωρών. Φυσικά, σε αυτή τη θεματική διαβολή δεν συμμετέχουν όλε όλες οι χώρε του κόσμου. Θα πρέπει να τι εμπλέξουμε όσο μπορούμε. Και εσεί κυρίω οι ευρωβουλευτέ που έχετε πολλέ ε, επαφέ με τρίτες χώρε, θα πρέπει να παίξετε σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει λοιπόν ε, να συνεργαστούμε με χώρε που έχουν την ίδια άποψη στα πλαίσια αυτή τη διπλωματία, να δημιουργήσουμε ε, συμμαχίε, γέφυρε για να αποφύγουμε του κατακαιρματισμού στο μέλλον. Από πλευρά μα θα πρέπει επίση να είμαστε ενωμένοι ε, είναι προφανές. Ο λόγος, όπως συζητήσαμε και στο παρελθόν, ε, που καταφέραμε να παίξουμε τόσο σημαντικό ρόλο, είναι ότι είχαμε μια πολύ καλή ε, ενωσιακή συμμετοχή, στην πούμε έτσι, στα πλαίσια της προετοιμασίας των θεματικών διαβουλεύσεων που γίνονται με τους δύο διευκολυντές, τον Μεξικανό και τον Σουηδό όπου τα κράτη-μέλη ε, παίρνουν το λόγο και η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει το λόγο. Και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό και θα πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Γιατί ακόμα κι αν δεν το συνειδητοποιούμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σαφές ότι όταν είμαστε στην Νέα Υόρκη, στη Γενέβη, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη, 28 χώρες δηλαδή, νομίζω ότι κάνουμε τη διαφορά. Δημιουργεί μια αίσθηση ε, και να μην την υποτιμούμε. Και ελπίζω να χρησιμοποιήσουμε αυτή την στήριξη που προσδίνουμε στις, στους στόχους κυρίας Άρμπουρ. Λοιπόν, ο συντονισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό σε αυτό το γύρο. Νομίζω, το ανέφερα και την τελευταία φορά το εξή, ότι για αυτέ τι θεματικέ διαβουλεύσει τα κοινοβούλια μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο, δηλαδή να δώσουν και αυτά τη δική του συνεισφορά και άποψη. Πολύ ωραία. Ε, θα πρέπει να έχουμε το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον για να δούμε τι θα γίνει μετά. Ε, αρχίζει, καθώς θα διαμορφώνεται το πράγμα, θα βλέπουμε τα θέματα, τα θέματα τα οποία σκιαγράφησε η κυρία Άρμπορ, ε, θα δούμε πώς θα τα προωθήσουμε με πρακτικό τρόπο, ούτω ώστε να έχουμε ένα σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης της ανθρώπινης κινητικότητας. Ε, έλευση, φυσικά, και στον ΟΗΕ και σε άλλα βήματα. Δουλεύουμε για τη μετανάστευση επί πολλά χρόνια. Αλλά το θέμα είναι να κάνουμε ένα ποιοτικό άλμα, ε, ούτω ώστε να υπάρξει αυτή η διακυβέρνηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κυρία Μουγκερίνη είναι πολύ υπέρ αυτή τη ιδέα και σίγουρα θα το πει στο, στη Σύνοδο αυτό το θέμα. Είναι τμήμα του, του αφηγήματό τη. Πάντα μιλάει για την ε, τεράστια σημασία, τις αξίες και την ευθύνη ε, που έχουμε σε επίπεδο που έχει μάλλον ο ΙΕΛ, ο οποίο είναι στον πυρήνα αυτή τη διαδικασία. Εμεί, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουμε να συνεισφέρουμε και να υποστηρίξουμε τη δουλειά που κάνει ο ΙΕΛ όσο μπορούμε, ούτω ώστε να είναι επιτυχής μέχρι τα τέλη του 2018 και να έχουμε ένα ποιοτικό σύμφωνο, φιλόδοξο, που να είναι κάτι παραπάνω από μια μοναδική εκδήλωση που σταματάει εκεί. Οι προσδοκίες είναι υψηλές, αλλά με τη συνεργασία και την στήριξη νομίζω ότι θα καταφέρουμε να τελεσφορήσουμε στις προσπάθειες. Ευχαριστώ. Πριν πάμε στη συζήτηση, για θα πρέπει να ξεκινήσουμε, να ακούσουμε την Τζένια Μπρόση για τον Διεθνή Οργανισμό για την Μετανάστευση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θαυμάσια επαφή που είχατε με την υπηρεσία στις Βρυξέλλες θα σας, ακούσουμε, λοιπόν και μετά θα περάσουμε στη ζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να παραβρεθώ εδώ και να μιλήσω με την κυρία Άρμπορ και με τη Λότε. Μας τιμά και εμένα ιδιαίτερα το ότι μπορούμε να σας αναφέρουμε κάποιες παρατηρήσεις μας. Για να δούμε γενικά ποια είναι τα κύρια θέματα που θα πρέπει να συζητήσουμε καθοδόν. Θα ήθελα να συμμεριστούμε κάποιες ε, απόψεις με τους εταίρους μας σε σχέση με την κατάσταση στο μεταναστευτικό και την αυξανόμενη ροή προς την Ευρώπη και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει αυτό το Global Compact Process προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή για να διαχειριστεί την τωρινή κατάσταση. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το εξή. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες βέβαια στο εσωτερικό της Ένωσης για συναπόφαση κάποια μια κλειδί. Ροές, μετανάστευση γενικότερα, θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης καμιά φορά δεν ομονοούν με τις χώρες μέλη ή κάποιες χώρες μέλη και καταβάλλεται μια προσπάθεια εδώ και καιρό ώστε να υπάρξει έτσι μια ενότητα όσον αφορά όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το θέμα και στα πλαίσια αυτού του περίπλοκου κόσμου μη σύμπαντος που αποτελεί Έχουμε την ε, δήλωση της Νέας Υόρκης, διακήρυξη συγγνώμη, που υιοθέτησαν οι χώρες του ΙΕ χώρες μέλη του ΙΕ κατά συνέπεια της Ένωσης και προσφέρει μια βασική αρχή, συμπεφωνημένη δηλαδή, που μπορεί να βοηθήσει και την Ένωση αλλά και τις χώρες της ώστε να προσπαθήσουν να διαχειριστούν και να επιλύσουν κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τώρα. Και μην ξεχνάμε ότι η διακήρυξη της Νέας Υόρκης και η περσινή διάσκεψη απετέλεσαν ιστορικές στιγμές γιατί όπως ξέρετε στον ΟΗΕ είχε γίνει προσπάθεια επανειλημμένως για συνέβρεση ηγετών παγκοσμίω για να συζητήσουν για αυτά τα θέματα αλλά δεν συνέβη επειδή κάποιε χώρε δεν το επιθυμούσαν αυτό, δεν το ήθελαν μέχρι πέρσι. Αυτό είναι λοιπόν ένα ορόσημο. Η διακήρυξη της Νέας Υόρκης είναι ένα ορόσημο και το ακούσαμε προηγουμένως. Είναι πολύ σημαντικό θέμα η διακήρυξη. Εμείς που εργαζόμαστε σε αυτό το τομέα θεωρούμε ότι κάθε μετανάστης ανεξάρτητα διοικητικής ε, κατάστασης καθεστώτος πρέπει να προστατεύεται αυτός και τα δικαιώματά του. Αλλά αυτό δεν έγινε αυτομάτως. Οπότε η πρώτη ευκαιρία για την Ένωση είναι ακριβώς αυτό το σημείο κίνησης αυτής της διαδικασίας που αποτελεί μια βελτίωση σε σχέση με τη διαχείριση της πολιτικής της μετανάστευσης, ώστε αυτή να γίνει πιο συνεπής σε σχέση με αυτά που έχουν αποφασιστεί σε επίπεδο μεμονωμένων χωρών μελών της Ένωσης ή ενωσιακό σε σχέση με διάφορες πτυχές μετανάστευσης. Κάποια άλλα ζητήματα που νομίζω ότι αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την Ένωση είναι καταρχάς ότι μετά από κάποια χρόνια και έχοντας επικεντρωθεί σε αυτά που γινόταν στα εξωτερικά σύνορα, αφήξεις, τι κάνουμε και όπως είπε σωστά η Λότε, όλα αυτά έχουν φύγει πια από το καθημερινό λεξιλόγιο κάποιων χωρών της ένωση, όχι όλων. Τώρα με αυτή τη δικασία η Ένωση έχει τη δυνατότητα να δει σφαιρικότερα τη μετανάστευση. Πέραν δηλαδή από τι προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα. Και αυτό είναι σημαντικό για να έχουμε μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση. Είναι σημαντικό ακριβώς για να αποτιμήσουμε και τον παγκόσμιο αντίκτυπο της κινητικότητα και να περάσουμε από απαντήσεις που όσον αφορά τις πολιτικές στην Ένωση ήταν περισσότερο εκτακτής ανάγκης, δηλαδή βραχυπρόθεσμες θέματα ημερών, χωρίς όμως να υπάρχει μια προσέγγιση μακρόπνοη. Οπότε και πάλι με αυτές τις συζητήσεις και με αυτή τη δικασία έτσι όπως έχει δομηθεί θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για την Ένωση για να προχωρήσει ακριβώς προς μια σφαιρικότερη προσέγγιση. Δεν ξέρω έχω χρόνο ακόμα να πω και το εξή. Ένα άλλο σημείο που είναι μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση είναι ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε στα πλαίσια αυτή τη διαδικασία global, global Compact Process, ώστε να βελτιωθεί, να βελτιωθεί η ίδια η ενότητα της Ένωσης στα πλαίσια της πολιτικής μετανάστευσης. Δηλαδή, μια διαδικασία που όπως είδαμε στην προετοιμασία της ε, διάσκεψης κορυφής πέρσι ενθαρρύνεται να δουλέψει με πιο ενωμένο τρόπο, να έχει πιο ενωτικές θέσεις ώστε να βελτιωθεί και το επίπεδο συνεργασίας και ο κοινό χαρακτήρας των πολιτικών στο εσωτερικό του χρόνου της Ένωσης που μέχρι τώρα κατά κάποιο τρόπο ήταν κατακαιρματισμένε, επειδή κάθε χώρα μέλο τη Ένωση είχε τη δική της πολιτική για πολλά αυτά τα ζητήματα. Οπότε αυτή η διαδικασία και πάλι θα αποτελέσει μια οθήση, μια επιπλέον οθήση, ώστε η Ένωση και τα θεσμικά τη όργανα να καταβάλουν περισσότερε προσπάθειε προ μια ενιαία δράση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα και ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε Ιδίω την προσκεκλημένη μας ε, Λουίζα Άρμπορ και για την συνεισφορά τη στη συζήτηση χθε. Τα περισσότερα μέλη της Επιτροπής ε, σας παρακολούθησαν και χθες. Ε, η, την ομιλία μάλιστα συνάδελφοι την έχουμε, είναι εξαιρετική αν τη θέλετε. θα ακούσουμε τώρα κάποιες παρεμβάσεις από ευρωβουλευτές και στη συνέχεια θα σας ξαναδώσω το λόγο. Η κυρία Ζήπελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τους ομιλητές. Εκτιμώ πολύ το γεγονός ότι στις παρεμβάσεις σας εισηγητικά προσπαθήσατε να εστιάσετε σε κάποια θετικά σημάδια που βλέπουμε στον τομέα της μετανάστευσης και της συνεργασίας. Παρ' όλα αυτά, Και ερχόμενοι στο θέμα της διακήρυξης, πρέπει να πω ότι έχουμε δει πολλές διακήρυξεις και θετικότατες μάλιστα για τη μετανάστευση. Στην πράξη όμως τα πράγματα δεν είναι πάντοτε τόσο θετικά. Θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Δεν μπορεί κανείς φυσικά να πει ε, τίποτα εναντίον ε, της, του ελέγχου των, ε, των συνόρων. Φυσικά και είναι απαραίτητο το να υπάρχει προστασία των συνόρων. Ωστόσο, όταν στο τομέα τη μετανάστευση επικεντρωνόμαστε μόνο στον έλεγχο των συνόρων και την καταστολή, τότε καθιστούμε το ταξίδι των μεταναστών που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τι αστείε του πιο δύσκολο, πιο επικίνδυνο και στην ουσία ε, μια τέτοια στάση συμφέρει μόνο τους διακινητές. Ε, πολλές φορές μάλιστα ακούμε απόψεις που λένε ότι ο έλεγχος των συνάρων συνόρων είναι σημαντικός γιατί θα μπορούσε να, να μειώσουμε τους ανθρώπους, τους μετανάστες. Δεν μειώνονται οι μετανάστες. Μειώνονται αυτοί που έρχονται στις χώρες μας, στα σύνορά μας. Εν πάση περιπτώσει, θετική εξέλιξη θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει ε, μια κάπως μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε αυτό που είχαμε αποκαλέσει εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο μια ολιστική προσέγγιση. Να αναγνωριστεί δηλαδή ότι χρειάζεται διαχείριση της μετανάστευσης, ότι αντιμετωπίζονται προκλήσεις ε, στην Ευρώπη όσον αφορά την υποδοχή και τη φιλοξενία των προσφύγων, αλλά υπάρχουν προκλήσεις και εκτός Ευρώπης. Ε, που ε, αφορούν ιδίως τα ριζικά αίτια της μετανάστευσης και πρέπει να δοθούν λύσεις και στους δύο τομείς. Για να επανέλθω τώρα στο διεθνές επίπεδο υπάρχει μια μικρή χαραμάδα ελπίδας στην οποία εγώ θα ήθελα να εστιάσουμε για να γίνει πραγματικότητα. Πολλές φορές ε, ακούγονται αλληλοκατηγορίες. Ποιος πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα, Ποιος πρέπει να ε, αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση ως προς τη διαχείριση της μετανάστευσης. Κατά τη γνώμη μου η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτή τη μεγάλη πρόκληση της μετανάστευσης. Ε, έχει βεβαίως ορισμένες ε, από τις ευθύνες για τα ριζικά αίτια. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε ότι να δούμε τι θα κάνουν οι διεθνείς ε, οργανισμοί. Αντιθέτως, πρέπει τα κράτη-μέλη της Ένωσης να αποτελέσουν παραδείγματα προς μίμηση για τη διαχείριση της μετανάστευσης τόσο εσωτερικά όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μόνο τότε μπορούμε να στραφούμε σε άλλες χώρες στο διεθνές στερέωμα και να πούμε «Είδατε, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, το κάναμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» Διαχειριζόμαστε την μετανάστευση και σα καλούμε να κάνετε το ίδιο. Δεν βλέπω να υπάρχει μια τέτοια εξέλιξη, μια τέτοια κίνηση αυτή τη στιγμή. Αυτό όμω θα ήθελα εγώ να δω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να κρύβεται πίσω από διεθνεί οργανισμού. Αντιθέτω, να κάνει εκείνη το πρώτο βήμα να επανέλθει δηλαδή σε μια ολιστική προσέγγιση, να κάνει αυτή την, το, το πρώτο βήμα, να, να αποτελέσει εκείνη την αφετηρία για μια νέα διαχείριση μετανάστευση και από εκεί και πέρα να καλέσει και τους άλλους να κάνουν το ίδιο. Η κυρία Δεοζιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπατε κι εσείς, ορισμένοι από εμά συμμετείχαμε στη χθεσινή διάσκεψη. Κυρία Άρμπορ, η παρέμβασή σας ήταν ε, μία πνοή φρέσκου αέρα ε, μετά από διάφορες παρεμβάσεις που άκουσα. Σημερίζομαι συμμερίζομαι σε μεγάλο βαθμό τα λεγόμενά σας. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα, ούτως ώστε να στηριχθούμε σε γεγονότα. Και μάλιστα θέλω να υπενθυμίσω και μερικά. Υπάρχουν 244 εκατομμύρια διεθνών μεταναστών σε όλο τον πλανήτη. Είναι το 3,3 ε, του πληθυσμού σήμερα και ήταν το 2,9 ε, του πληθυσμού το 1990. Αυξήθηκε, αλλά σε σχέση με την παγκόσμια κινητικότητα δεν αυξήθηκε τόσο δραματικά. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το πούμε πολλές φορές, έτσι και να το τονίσουμε. Δεύτερο στοιχείο, που με εκπλήσει κιόλας. Ξεχνάμε να βάλουμε ε, στη συζήτηση αυτή τη θέση των Ευρωπαίων ε, μεταναστών. Υπάρχουν 60 εκατομμύρια διεθνών μεταναστών που είναι Ευρωπαίοι. Για μία Ήπειρο ε, που έχει 500 εκατομμύρια κατοίκους. Υπάρχουν 34 εκατομμύρια Αφρικανών μεταναστών για μια Ήπειρο που έχει 1,2 δισεκατομμύρια άτομα. Και 80% των διεθνών μεταναστών είναι μετανάστες ενδοαφρικανοί, δηλαδή από μια χώρα της Αφρικής σε μια άλλη. Εάν θέλουμε λοιπόν ε, να θέσουμε τα κράτη μας ενώπιον των ευθυνών τους, θα πρέπει όλα αυτά να τα βάλουμε στο παγκόσμιο πλαίσιο. Και όταν λέτε ας στηριχθούμε στα γεγονότα, θα ήθελα να τα θέσουμε όλα αυτά με ένα τέτοιο τρόπο, ούτω ώστε να έχουμε ένα βλέμμα, μια ματιά, ε, λιγότερο δυτικό, κεντρικό και να έχουμε μια έτσι πιο παγκόσμια θεώρηση της μετανάστευσης. Δεύτερον, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε για το πόσο σημαντικό είναι να πούμε ότι όλοι οι μετανάστες ε, έχουν δικαιώματα. Ανά, ανεξάρτητα από την κατάστασή τους. Έχουμε τρεις εκθέσεις όπου μιλήσαμε για αυτό το θέμα. Το ένα το δικό μου για τη μετανάστευση και τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες. Υπενθυμήθηκε και στην ε, έκθεση Μετσόλα και Εγγέμ, ε, καθώς και στην ε, έκθεση Δίας Δεμέρα Βαλενσιάνου. Υπενθυμίζουμε αυτό το θέμα και υπενθυμίζουμε την ανάγκη τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπογράψουν τη Διεθνή Σύμβαση των μεταναστών ε, εργαζομένων και των οικογενειών τους. Και αυτό θα πρέπει να μπει ψηλά στην ατζέντα μας. Πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να δούμε μέσα σε μια προοπτική και μέσα σε ένα πλαίσιο. Επίσης το θέμα της μετανάστευσης να το βάλουμε ε, όχι μόνο σε πρόβλημα, αλλά να το δούμε συνολικά. Το έχω πει και θα το ξαναπώ τώρα υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια άτομα τα οποία κάθε χρόνο έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υπήκοοι τρίτων χωρών με θεωρήσεις ε, μακράς διάρκειας χωρίς να μιλήσουμε για την εντοκινοτική κινητικότητα, έτσι, χώρια από αυτήν. Από αυτά τα άτομα υπάρχουν 500 Ουκρανοί, 250.000 250 ε, ε, Ινδιάνοι, 250.000 ε, Κινέζοι και άλλοι τόσοι Αμερικανοί. Αυτά τα νούμερα πού θα τα πούμε για να δείξουμε ότι στην πραγματικότητα η μετανάστευση ε, είναι πολύ πιο περίπλοκη. Δεν υπάρχει μόνο η προβληματική μετανάστευση. Είναι η πραγματικότητα και θα σταματήσω εδώ για να μην ε, μακρηγορήσω. Είναι το πώς εμείς βλέπουμε το θέμα, ε, η δική μας η θεώρηση, η δική μας η ματιά. Πώς να το πω. Έχουμε μια ματιά όλο και πιο ρατσιστική και ξενόφοβη θα έλεγα. Το θέμα των μεταναστών που προτάσουμε ποιο είναι. Είναι οι μετανάστες που έρχονται από τον Νότο. Αυτοί μας ενοχλούν, όχι εμένα, άλλους. Ε, δημιουργούν πρόβλημα στους κυβερνώντες μας. Λοιπόν, πρέπει όλα αυτά τα νούμερα να τα πούμε. Εάν θέλουμε να βγούμε από το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, όλα αυτά τα νούμερα να τα αναφέρουμε. Γιατί και αυτά είναι στοιχεία. Ε, είναι πολύ πιο πλατή το πρόβλημα. Και αν δεν σταματούμε να λέμε τα ίδια και τα ίδια, θα έχουμε πρόβλημα. Θα ήθελα λοιπόν όλα αυτά να προτάσσονται στα διάφορα έγγραφα που ετοιμάζουμε. Γιατί νομίζω ότι επικεντρωνόμαστε υπερβολικά στην λαθρομετανάστευση και στους πρόσφυγες. Υπάρχει ένα, μια τεράστια μάζα ανθρώπων ε, που υποφελείται από την κινητικότητα. Την τελευταία φορά που ήρθατε να μας δείτε, τονίσατε λίγο περισσότερο αυτό το στοιχείο της κινητικότητας και θα ήθελα να μην το ξεχάσετε αυτή τη φορά. Ε, ε, μια χαρά θα πάμε με το χρόνο. Μην αγχώνεστε. Βλέπετε ε, ότι ως Καναδί είναι δίγλωση η προσκεκλημένη μας και δεν χρειάζεται διερμηνία. Η κυρία Τούνσταϊν που μάλιστα παρευρέθηκε στην ε, σύνοδο της Νέας Υόρκης ως μία από τις τρεις ε, ευρωβουλευτές που παρευρέθησαν εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ και με τις δύο συναδέλφους και με εντυπωσίασε και εμένα αυτή η εκδήλωση χθες. Χαίρομαι πολύ που έχουμε την ε, ικανότητα να διοργανώνουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Ήταν πολύ διπλωματικός ο τρόπος που διατυπώσατε το, το θέμα της αντιμετώπισης ε, του κατακαιρματισμού των πολιτικών μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ ε, υψηλός αυτός ο κατακαιρματισμός, αν και, ε, και, και πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα σε πολλούς τομείς. Νομίζω ότι σε έναν βαθμό ε, μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτόν τον κατακαιρματισμό των πολιτικών για τη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν αποκτήσουμε και μια καλύτερη επικοινωνιακή πολιτική. Και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορούμε να το κάνουμε τόσο ε, ε, ε, εσωτερικά, αλλά και με τα άλλα κράτη. Και με τα άλλα κράτη. Ε, όταν μιλούμε για επικοινωνιακή πολιτική, η καλή διαχείριση των συνόρων είναι και μια ορθή επικοινωνική πολιτική που απαντά στους λαϊκιστές που μπλέκουν σκόπιμα και συνειδητά τους μετανάστες και τους πρόσφυγες με τους τρομοκράτες γιατί βασίζονται στον φόβο, προκαλούν τον φόβο των πολιτών και ο φόβος ξέρετε είναι κάτι που ε, διαχέεται πολύ γρήγορα και εύκολα. Πέραν λοιπόν από τον κατακαιρματισμό όσον αφορά τις πολιτικές, όταν ακούω ε, πώς λειτουργούν οι αρχές ελέγχου των συνόρων σε διάφορες χώρες, στις επισκέψεις μου αλλά και στις συνομιλίες μου ε, που είχα με ανθρώπους που αποφασίζουν σχετικά με το καθεστώς των μεταναστών που έρχονται στην Ευρώπη. Είναι τόσο διαφορετικές οι, οι πρακτικές που ακολουθούνται και μάλιστα ορισμένες φορές τόσο άδικες ε, όταν ακούω ε, για ανθρώπους που ρωτούν, για, που, θέτουν ερωτήσεις ε, για τις πόλεις ε, και, και την κατάσταση που επικρατεί στην ε, ε, στην ε, χώρα προέλευση τους όταν οι ίδιοι μετανάστες αντιμετωπίζουν και την αμφιβολία των αρχών δεν τους πιστεύουν πολλές φορές αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν δαπανίσουμε περισσότερα χρήματα περισσότερο χρόνο ε, περισσότερες προσπάθειες για να επικοινωνήσουμε τις δικές μα πολιτικέ για να αντιμετωπίσουμε εκείνου που διασπείρουν τον φόβο νομίζω ότι θα ήταν ένα τρόπο. Ε, για να οικοδομήσουμε μια κοινή πολιτική, να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα, μεγαλύτερη εμπλοκή και συμμετοχή των πολιτών μας ε, στις, ε, στους κοινούς στόχους και σκοπούς που έχουμε εδώ στην Ήπειρό μας. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Βίνμπεργκ. Ευχαριστώ, διακήρυξη της Νέας Υόρκης. Παγκόσμια ελεγγύη. Ωραία ακούγεται. Αλλά νομίζω επιφέρει και μια ευθύνη και κάτι το οποίο ακούγεται θετικά. Όμως ας δείξουμε μια ματιά στο εσωτερικό της Ένωσης και τι προσπαθήσαμε να κάνουμε εκεί τα τελευταία χρόνια με την ε, αλληλεγγύη μας. Αυτή η ελεγγύη σε θελούσια βάση καλή είναι θεωρητικά, αλλά δεν είναι αποτελεσματική. Και τώρα έχουμε μια υποχρεωτική ελεγγύη στο εσωτερικό της Ένωσης. Γιατί αυτό ακριβώς θα γίνει με διάφορα κονδύλια, τα οποία όμως δεν θα δίδονται αν δεν τηρηθούν κριτήρια κατανομής. Οπότε κατά κάποιο τρόπο είναι επιβεβαιωμένη αυτή η αλληλεγγύη. Η κυρία Άρμπορ μίλησε για εναλλακτικέ λύσεις όσον αφορά αυτούς που είναι απροστάτευτοι. Βεβαίω η πλειοψηφία των μεταναστών, το 70% αυτών που καταφθάνουν στην Ευρώπη, είναι οικονομικοί μετανάστες. Εσείς ας πούμε Μήπως έχετε κατά νου αυτούς που ενδεχομένως δεν χρειάζονται προστασία υπό την έννοια δηλαδή ότι θέλουμε να πούμε βοήθεια για την έρευνά τους ή για κάτι τέτοιο. Έχουμε την μπλε κάρτα στην Ένωση. Μέχρι 3.000 άτομα μπορούμε να δεχτούμε αιτησίως. Ε, οπότε εσείς ποιες εναλλακτικές έχετε κατά νου για να καταλάβω. Επιπλέον να πω έχουμε αυτά τα 6-7 εκατομμύρια άτομα τα οποία βρίσκονται στην Αφρική και τα οποία θα ήθελα να μεταναστεύσουν. Είναι άτομα τα οποία προσπαθούν να φτάσουν από την Αφρική στην ε, Ευρώπη. Η πλειοψηφία όμως των χωρών προέλευσης αυτό το μεταναστών, σε ποια κατάσταση θα είναι σε 5, 10, 50 χρόνια, αν λάβουμε υπόψη μα το συνολικό αριθμό αυτών που θέλουν να καταστάσουν εδώ στην Ευρώπη. Τι γίνεται. Ευχαριστώ. Η οποία χθε μίλησε για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι μίλησε στην τελική φάση της διάσκεψης. Δεν ξέρω αν είχες φύγει τότε. Μπορείς να επαναλάβεις κάποια από αυτά που είπες χθε, όχι όλα. Ε, ο, ανεβάζει τον πύχη τώρα. Προσπαθούσα να συνέλθω μετά την προηγούμενη παρέμβαση. Ε, γιατί εγώ έχω μία άποψη για τους Σκανδιναβούς. Είναι γνωστή για την αλληλεγγύη τους. Όταν τους ακούω να μιλάνε λοιπόν για αναγκαστική αλληλεγγύη, που, ε, αλληλεγγύη δηλαδή που επιβάλλεται άνωθεν, εκπλήσει. Μία παρατήρηση και μία ερώτηση. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, αν κοιτάξετε τα νούμερα των, των ανθρώπων που έρχονται στην Ευρώπη, που ήρθαν, ας πούμε, το τελευταίο χρόνο, 1,5 χρόνο, πολλοί κόσμος. Και όμω είναι 0,2 με 0,3 του πληθυσμού. Εάν θεωρούμε ότι η ταυτότητά μα και ο τρόπος ζωής μας ε, απειλείται από το 0,3% του πληθυσμού, τότε η ταυτότητά μα δεν είναι και τόσο ισχύρη, έτσι. Μήπω πρέπει να το σκεφτούμε λιγάκι αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, υπάρχει μια τάση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να είναι πολύ πιο συγκεκριμένη. Τα κράτη-μέλη και οι κυβερνήσει, το Συμβούλιο, δηλαδή αυτοί που συνεδριάζουν τώρα, 28 άτομα, αυτοί είναι εντελώς ανίκανοι να συμφωνήσουν για το θέμα. Είναι ντροπή. Που βλέπουμε πόσο πολύ, πολύ πιο εύκολα τα καταφέρουν να συμφωνήσουν να με δικτάτορε παρά να συμφωνήσουν οι αρχηγοί μεταξύ του. Ε, Επομένω, λοιπόν, εξάγουμε το πρόβλημα, επειδή δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για μια δική μα πολιτική. Το εξάγουμε στην Τουρκία, στην Ερυθρέα, στη, στο Σουδάν, το εξάγουμε στη Λιβύη και σε άλλα λαμπρά παραδείγματα δημοκρατία και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Συμβούλιο, οι αρχηγοί μάλλον των κυβερνήσεων και μερικέ φορέ με τη συνοχή τη Κομισιόν, πρέπει να πω, έχουν την τάση να εκφεύγουν από το πλαίσιο των ευρωπαϊκών συνθήκων. Βολικότατο, γιατί τα, δεν ισχύουν τότε τα πρότυπα, δεν υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος, ούτε ενδικά μέσα, ούτε λογοδοσία, τίποτα. Επομένως, οι αρχηγοί, οι και κυβερνήσεων και η εθνική πολιτική ε, προτεμούν να διασπείρουν φόβο και τρομακτικέ ιστορίε ότι θα μα πλημμυρίσουν οι τρομακτικοί αυτοί ξένοι, θα εισβάλλουν σε εμά, αντί και τους λένε «Α, κοιτάξτε τι κάνουμε» είναι ε, υποδοχή ε, στην περιφερειά τους. Γιατί ο κόσμος προστιμάει να είναι κοντά στο σπίτι του, του ζήσει και λίγα λεφτά και είναι μια χαρά. Έτσι. Πεστε μου εσείς τώρα. Γιατί ακούω τους αρχηγούς μας να λένε ότι αυτά τα συστήματα με την Τουρκία Φερρυπίν ή το σύστημα το οποίο δεν το διαφημίζουμε, το να δώσουμε 90 εκατομμύρια στην ε, Λιβική ακτοφυλακή, 100 εκατομμύρια σε ε, στους δικτάτορες της Ερυθρέας και του Σουδάν, είναι τέλεια, μεγάλη επιτυχία. Πέστε μας εσείς, όταν μιλάτε στους πολίτες, στους ε, εκλογείς, ε, να μας πούν τι σημαίνει αυτή η υποδοχή στην περιοχή. Ε, εσείς θεωρείτε ότι αυτό είναι μια καταπληκτική επιτυχία. Πέστε μας αυτό το πράγμα. Η υποδοχή στη συγκεκριμένη περιοχή, στην περιφέρεια, την οποία προέρχονται. Έχουμε πολλούς ενδιαφέροντες προσκεκλημένους συχνά, αλλά όχι ε, τέτοιους που να μας δίνουν αυτήν την οπτική του ΟΗΕ, του Καναδά, όσον αφορά αυτές τις πολιτικές ενσωμάτωσης, ένταξης, όπως αυτές οι πολιτικές που μας παρουσιάσατε χτες. Θέλω λοιπόν να θέσω αυτό το ερώτημα της προοπτικής. Εγώ δεν είναι γνωστό. Ε, ήρθα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ινδία. Ξέρω λοιπόν, έχω βιώσει ε, ποια είναι η αντίσταση που προβάλλεται πολλές φορές σε ανθρώπους ε, που δεν είναι λευκοί, που έρχονται στην Ευρώπη από άλλες χώρες και υπήρους. Η χθεσινή σας ομιλία είχε έναν πολύ έντονο πολιτικό και ειλικρινή χαρακτήρα. Οι άνθρωποι λοιπόν προβάλλουν αντίσταση στη διαφορετικότητα. Αυτό είναι, είναι γεγονός. Αυτό που βλέπουμε στον Καναδά είναι ότι προφανώς τα πράγματα δεν είναι τέλεια. Καμία δυτική χώρα δεν είναι τέλεια. Ε, ε, ε, είμαστε τέλειοι, λέει η ομιλήτρια. Όχι, το φαντάστηκα ότι θα τα λέγατε. Εν πάση περιπτώσει, είναι, είναι, είναι, αγγίζει την τελειότητα. Αυτό που όμως ε, με ενδιαφέρει εμένα είναι πώς καταφέρατε να αλλάξετε την, την οτροπία των ανθρώπων. Γιατί εδώ βλέπετε και, στην, και από αυτό που είπε η κυρία Ίντβελ, ότι στην Ευρώπη κυριαρχεί η άποψη ότι είμαστε μια πολύ μικρή ήπειρος, ε, στην, ε, στις βαλτικές χώρες δεν υπάρχουν, πάρα πολύ, δεν υπάρχουν πολλοί μετανάστες, ενώ στη Δυτική Ευρώπη, στις πόλεις της Δυτικής Ευρώπης μας έχουν πνίξει μετανάστες ε, ε και ότι αντιμετωπίζουμε αυτές τις πιέσεις, πληθυσμιακές πιέσεις, θρησκευτικού χαρακτήρα, εθνοτικού χαρακτήρα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, ως δυτική χώρα, τι μέτρα μπορεί να λάβει κανείς για να, αλλάξει αυτή, να αλλάξουν αυτές οι αντιλήψεις, για να αλλάξει η νοοτροπία, ώστε να κατανοήσουν οι άνθρωποι ότι η μετανάστευση είναι και ένα στοιχείο απαραίτητο και αναγκαίο στη σύγχρονη εποχή. Ε, τα, τα, μέτρα, τα κοινά μέτρα διαχείρισης της μετανάστευσης, της νόμιμης μετανάστευσης, δεν είναι πολλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την μπλε κάρτα, στην οποία προβάλλουν τεράστια αντίσταση όμως τα κράτη-μέλη και είναι σχεδόν μόνο αυτό. Παρότι λοιπόν πολλοί από εμά ε, δουλεύουμε πάνω σε, σε αυτά τα προοδευτικά θέματα, αυτό που μας δυσκολεύει είναι τα μέτρα ελέγχου που βεβαίως πολλοί θέλουν. Το ερώτημα μου είναι, σε μια χώρα όπως ο Καναδάς γνωρίζουμε ότι η αντίληψη που έχει επιτευχθεί είναι πιο ισορροπημένη, όχι μόνο απέναντι στην λευκή μετανάστευση, αλλά και από χώρες όπου το χρώμα του δέρματος των ανθρώπων είναι πιο σκούρο. Θέλω λοιπόν να μου πείτε εσείς πόσο ενεργά πρέπει οι κυβερνήσεις ε, οι κρατικές υπηρεσίες, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, δεν ξέρω ποιος ακριβώς τελικά τίθεται επικεφαλής, τι πρέπει εν πάση περιπτώσει να κάνουν για να ε, χαραχτεί μια τέτοια πορεία. Αυτά από μένα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος που θα θέλει το λόγο. Ήρθε μόλις η Μπάρμπαρα. Εν πάση περιπτώσει θα κάνουμε και ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Θα κάνουμε και δεύτερο, αν θέλετε, αν υπάρχουν και άλλα ε, ερωτήματα για να τα θέσετε. Κατερίνα, Κατερίνα Κινίτσι. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι επίσης ε, δικαστής και είμαι ε, και εγώ από αυτούς που πιστεύουν ότι είμαστε τέλειοι. Πλάκα κάνω. Ε, είμαι δικαστής λοιπόν και αντιμε... έχω μια τέτοια εμπειρία. Ε, προέρχομαι από μια χώρα, την Ιταλία, η οποία, ειδικά στην Σικελία, γιατί εγώ είμαι Σικελή, Μία πρακτική υποδοχής ε, ε, που είναι, ανάγεται στο παρελθόν, στο απότατο παρελθόν. Από τη Σικελία πέρασαν πάρα πολλοί λαοί, φυλές. Έχουμε αυτή την ε, ιδέα, την παράδοση της υποδοχής. Και την εκδηλώνουμε τώρα απέναντι στους μετανάστες που φτάνουν στις ακτές μας. Είμαστε στην, στην Μεσόγειο και φτάνουμε με δραματικό τρόπο δυστυχώς με αυτά τα σκάφη, με αυτές τις βάρκες, άτομα τα οποία προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες, φεύγουν από διώξεις, από συνθήκες ζωής άνθρωπες και διασχίζουν τη Μεσόγειο, κάνουν αυτό το ταξίδι της απελπισίας, έτσι το λέω, παρά το ταξίδι της ελπίδας, γιατί ε, η ελπίδα είναι ότι θα βρεις ε, συνθήκες ζωής ε, ανθρώπινες, αλλά αντιμετωπίζουν τη φρίκη. Εμείς κάναμε μια τεράστια προσπάθεια λοιπόν στη χώρα μου, μαζί με την εθνική κυβέρνηση, τις τοπικές αρχές, ε, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τους ίδιους τους πολίτες που ήταν έτοιμοι να υποδεχτούν, να χρησιμοποιήσουν από εκείνου τους πόρους και να κινητοποιηθούν όχι μόνο τη στιγμή της άφηξης των μεταναστών, τη στιγμή που υπάρχει κατεπίγουσα ανάγκη, αλλά να ξεκινήσουν μια διαδικασία ένταξης. Εγώ παρακολουθώ κυρίως τους ανήλικους, τους ασυνόδευτους ανήλικους Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από τη χώρα μου, πρέπει να σας πω. Λοιπόν, μπροστά σε χώρες τώρα, ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες υψώνουν τείχους, αν όχι φυσικούς, τουλάχιστον ε, με τα λόγια. Δεν ε, δηλώνουν διαθέσιμη για την υποδοχή, γι' αυτό λοιπόν ε, χάνω λίγο τον μπούσουλα απέναντι σε τέτοιες τάσεις. Διερωτώ με λοιπόν αυτό που διερωτάται και ο Κλοντ για το θέμα της στην περίπτωση της Αγγλίας. Αυτές οι χώρες που έχουν την ικανότητα, τη συνήθεια τέλος πάντων ε, του ανοίγματο. Όταν βλέπουμε χώρες που δεν έχουν αυτό το άνοιγμα σαν και εμάς, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εμπλέξουμε ακόμα περισσότερο τις άλλες χώρες. Εσείς είπατε προηγουμένως ότι μπορεί να είναι μια πρόκληση, μια δυσκολία, μπορεί να είναι και κάτι θετικό. Εγώ πιστεύω ότι κάθε πρόκληση μπορεί να μετασχηματιστεί σε κάτι θετικό, αν αντιμετωπίσουμε να την δούμε με το σωστό τρόπο. Νομίζω λοιπόν ότι σε πολιτικό επίπεδο, γενικά μιλάω τώρα έτσι, στην Ευρώπη, λείπει αυτή η ικανότητα να αντιμετωπίσουμε σωστά αυτό το θέμα. Γιατί και η Μπίργκετ αναφέρθηκε προηγουμένω στι ανησυχίε στου φόβου στο φόβο να, του να δεχθείς κάτι που είναι διαφορετικό από σένα. Ε, φοβόμαστε ότι θα εισβάλλουν στις μικρές μας πόλεις, ε, στη, στις θέσεις εργασίας μας κτλ. Πώς μπορούμε να τα ξεπεράσουμε σε πολιτικό επίπεδο αυτά, πώς μπορούμε εμείς οι χώρες οι οποίες ε, ξέραμε να το κάνουμε και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποδεχτούμε του ξένου, πώ μπορούμε να βοηθήσουμε, ούτω ώστε να δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια πολιτική αλληλεγγύη, που δεν είναι μια επιβεβλημένη αλληλεγγύη. Ε, το βλέπω με μεγάλη θλίψη, να ακούω με μεγάλη θλίψη τέτοιε δηλώσει και βλέπω με μεγάλη θλίψη αυτέ τι κυρώσει που επιβάλλουμε σε χώρε που δεν υποδέχονται. Εσείς λοιπόν που είσαστε από τον Καναδά, έχετε διαφορετική εμπειρία, τι προτάσεις μπορούμε να κάνουμε τόσο ώστε να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε μια σωστή, τη σωστή αντίδραση, να μετασχηματίσουμε το αρνητικό σε θετικό. Πώς γίνεται. Ευχαριστώ Κατερίνα. Ε, κοιτάξτε, το αδιέξοδο του Δουβλίνου είναι τεράστιο θέμα για μας στην Επιτροπή μας. Ένας μεγάλος φάκελος που έχει κολλήσει αυτή τη στιγμή. Η Μπάρμπαρα Σπινέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη. Καταρχάς που έφτασα τόσο αργά. Ε, ήμουν απασχολημένη. Ίσως το ερώτημά μου το ακούσατε ήδη λοιπόν, ή εν μέρη το ακούσατε. Ε, αφορά τις ε, συμφωνίες επαναπατρισμού, κυρίως στη Λιβύη. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, ως εκπρόσωπο του ΟΗΕ, είναι να μου πείτε τη θέση του ΟΗΕ για την κατάρτιση των ακτοφυλάκων της Λιβύης. Χθες ή προχθές, ο ειδικός εκπρόσωπος του ΟΗΕ ε, στη Λιβύη, ο Μάρτιν Κόμπλερ, είπε ότι είναι πάρα πολύ ανήσυχος από αυτή την απόφαση να δώσουμε κατάρτιση στην Λιβική ακτοφυλακή. Το είπε σε εμά, τους ε, ευρωβουλευτές. Και μας είπε, πηγαίνετε στο YouTube και θα δείτε πώς αντιμετωπίζουν οι Λίβοι ακτοφύλακες τους ε, μετανάστες. Ποιο αναλαμβάνει το καθήκον της διαχείρισης τους και της, ε, του επαναπατρισμού τους. τους ε, μετανάστες τους ε, ρίχνουν στη θάλασσα ή τους επαναπατρίζουν στη Λιβύη. Σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς συμβάσεις, προφανώς αυτά δεν γίνονται σεβαστά. Εγώ ανησυχώ, γιατί η Ιταλία ειδικά είναι στο πρώτο μέτωπο παροχής κατάρτισης τους Λίβιους ακτοφύλακες. Θα ήθελα να μου πείτε την γνώμη σας. Ζητώ συγγνώμη αν τέθηκε ήδη το ερώτημα. No, Barbara, there was some reference but not... Υπήρξε κάποια αναφορά. Αλλά όχι ακριβώς, όπως το ρώτησες. Τόσο πάντων υπάρχει και κάποιος από την υπηρεσία εξωτερικής δράσης σε περίπτωση που θέλουν να σχολιάσει για αυτά τα θέματα και τα ερωτήματα που ακούσαμε χθε. Ωραία. Να ζητήσω τώρα από Λιουζάρμπορ να σχολιάσει. Ευχαριστώ, λέει κύριε Άρμπορ. Ωραία. Ενδιαφέρουσε η απόψει που ακούσαμε και ανησυχία. Θα αναφερθώ σε ερωτήσει και μετά μια γενικότερη τοποθέτηση. Όταν πιέζει η κοινή γνώμη δεν είναι δύσκολο να χαράξει πολιτικές. Καμιά φορά είναι δύσκολο να βρει τα σωστά μέτρα βέβαια, αλλά είναι σχετικά εύκολο να χαράξει πολιτική. Αυτό που είναι πολύ δύσκολο αντίθετα είναι το να έχεις ένα επίπεδο ηγεσία που θα ηγείται όπως ακριβώς σημαίνει η λέξη. Δηλαδή να αφορά και την κοινή γνώμη αυτό. Δηλαδή να μπορούν να αποτιμήσουν κατά πόσο η πίεση τη κοινή γνώμη πηγαίνει στην λάθος κατεύθυνση. Και θα πρέπει δηλαδή να υποχωρεί σε μια παραπληροφορημένη ή κακώ πληροφορημένη κοινή γνώμη. Υπάρχουν επίση περιπτώσει όπου ο κόσμο έχει συγκεκριμένε απόψει με θανατική πηγή κτλ. Πολλά επίμαχα ζητήματα, αλλά τέλο πάντων, αν είστε ηγέτη πραγματικό, τότε θα πρέπει να ηγηθείτε. μέσω πυθούς και ηγεσία. Καμιά φορά όμως ο κόσμος δεν θέλει να πιστεί μέσω στοιχείων ή δεδομένων και να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Δεν να κάνουμε, έτσι είναι. Για το συγκεκριμένο ζήτημα τώρα, δεν νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε για μια βαθιά αλλαγή του αφηγήματος ώστε να κινητοποιηθεί η κοινή γνώμη στη σωστή κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή ακριβώς που απαιτεί η ηγεσία. Και η ηγεσία νομίζω θα αντιμετωπίσει την προτίμηση για αντιλήψεις σε, αντί για δεδομένα και αντίληψη αντί για γνώση. Οπότε δεν μπορούμε σε αυτές τις περιπτώσεις με συγκεκριμένα στοιχεία να εξειδικεύσουμε κάθε τομέα πολιτικών. Ας πούμε, αν δούμε ε, το κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε κάτι για τη μεταφορά με, για τη συγγνώμη, των επιδομάτων. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε απλά και μόνο. Είναι, δεν γίνεται, είναι αδύνατον. Και νομίζω ότι η Ευρώπη θα ήταν καλό και συνετό να καθοδηγείται ως χώρα προορισμού ως τόπος προορισμού, χώρος προορισμού. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Είναι η ιστορία, ο πολιτισμός, η κυριαρχία και η παράδοση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που οδήγησε σε, αυτόν. Οπότε, σε αυτό. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ κατάλληλη στιγμή τώρα να δούμε κατά πόσο αυτή η πρόκληση μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω αυτών των αρχών. Δεν μπορώ να σας κάνω μάθημα εγώ. Εσείς ξέρετε πώς θα λύσετε τα προβλήματά σας. Αλλά σε γενικέ γραμμές το ίδιο θα έλεγα στους φίλους μου στη Λατινική Αμερική που αντιμετωπίζουν μια δομή προκλήσεων που είναι τελείως διαφορετικές. Δηλαδή αυτές στις Φιλιππίνες, στην Ινδονησία, στο Μπαγκλαντές που εξάγουν μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού όπως συνήθως γυναίκες που πηγαίνουν στις χώρες του κόλπου όπου 80% εκεί των ε, μεταναστών είναι μετανάστες γυναίκες. Οπότε αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Δεν έχετε την πολυτέλεια να περιμένετε την κοινή γνώμη για να δράσετε. Εσείς πρέπει να δράσετε και να χαράξετε τις πολιτικές και που θα περάσουν μετά αυτές την κοινή γνώμη. Όλοι είμαστε και προϊόν της ιστορίας μας. Σήμερα σας μιλώ ως αξιωματούχος, ως διεθνής δημόσιος υπάλληλος όχι μόνο ως Καναδία, αλλά και εγώ είμαι προϊόν της ιστορίας μου. Όταν είπα ότι είμαστε σχεδόν τέλειοι, το νοούσα. Είμαστε σχεδόν. Δεν υπάρχει το απόλυτο εδώ. Και πρόσφατα λεγόταν όπου ο Καναδάς είναι η μοναδική χώρα του κόσμου μπορεί να κερδίσει εκλογές όντας υπέρμαχος της μετανάστευσης. Ε, δεν είναι ότι έχουμε κάποια ηθική ανωτερότητα σχέση με τους άλλους. Έχουμε μεγάλη επικράτεια, έχουμε ανάγκες ε, πληθυσμού, έχουμε μια μακροχρόνια παράδοση μετανάστευσης, πολλών μορφών μετανάστευσης και πρόσφατα για τους μετανάστες είχαμε μια πάρα πολύ επιτυχή εμπειρία με χορηγία τοπικών κοινοτήτων σε προγράμματα μετανάστευσης όπου δίδαμε κάποια χρήματα για να αποδεχτούν τοπικές κοινότητες, ε, Σύριους κυρίως μετανάστες, που αποδείχθηκε πάρα πολύ επιτυχής αυτή η προσπάθεια. Τώρα, εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή την πολυτέλεια να κάνουμε απ' έξω, από το εξωτερικό αυτής της πολιτικής επανεγκατάστασης. Δεν έρχονται κολυμπώντας βέβαια σε εμά οι μετανάστες. Είχαμε, έχουμε χερσαία συνορία τα οποία όμως δεν είχαν δεχτεί παραβιάσεις, παρόλο που έστω και αυτό αλλάζει λιγάκι. Είναι λοιπόν δύσκολο να συγκρίνει κανείς τη μια κατάσταση με την άλλη και να κάνει μαθήματα στον κόσμο για το τι πρέπει να κάνει και τι όχι. Εκεί που είμαστε λιγότερο τέλειοι, και να σας πω και μια ιστορία, είναι ενδιαφέρον. Είδαμε σε μια καναδική εφημερίδα την περσμένη εβδομάδα μια αναφορά ένα δημοσίευμα για κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις στον Καναδά, συγκεκριμένων και κάποιων μεγάλο ΜΚΟ στο ανθρωπιστικό τομέα, όπου μέσω των δημοσιογράφων ανακάλυψαν ότι κάποιοι που εργάζονται για τις επιχειρήσεις που καθαρίζουν τη νύχτα τα κτίρια, δηλαδή αυτοί που έρχονται στο χώρο εργασία, αφού φύγουν όλοι, καθαρίζουν του αλέτες, διάζουν τα καλάθια κτλ. Λοιπόν, αυτέ οι επιχειρήσει πληρώνανε αρκετά χρήματα σε αυτές τις επιχειρήσεις και μετά βρήκαν ότι αυτές οι επιχειρήσεις απασχολούσαν πολλούς παράνομους ή άτυπους μετανάστες που ήταν αντικείμενο κατάχρησης και αυθαιρεσιών. Βέβαια, δεν ξέρω ποια ήταν η αντίδραση του κοινού, αλλά το άρθρο αυτό δεν ρίχνε το αρθρο αυτο δεν έριχνε το φταίξιμο στους μετανάστες, αλλά σε όλους τους υπόλοιπους. Επειδή ακριβώς εμείς ήδη θα πρέπει να σταματήσουμε την ύπαρξη αυτού του είδους ε, καταχρήσεων ή αθαιρεσιών. Και ξέρω ότι αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Μου δόθηκαν κάποια στοιχεία τα οποία δεν γνώριζα να σας πω την αλήθεια, αλλά καταρχάς να δούμε τι γίνεται με αυτό το Global Compact δηλαδή για πρώτη φορά η παγκόσμια κοινότητα να συνεργαστεί για αυτό το θέμα και να προσπαθήσει να λύσει αυτό το ζήτημα με ορίζοντα δύο ετών. Αλλά εμεί θα πρέπει να έχουμε ένα ορίζοντα δεκαετιών όσον αφορά την ανθρώπινη κινητικότητα για να εξετάσουμε ακριβώ το πώ θα μπορούσαμε να εξοπλιστούμε καλύτερα για να το διαχειριστούμε. Και δεν θα είναι τέλεια τα πράγματα, έτσι. Πάντοτε θα έχουμε αυτού που κάνουν απάτε, αυτού που κάνουν αυθαιρεσίε, που αυθαιρετούν, αλλά εμείς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τις θετικές πηγές της μετανάστευσης και αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε στο ιστορικό πλαίσιο είναι ότι η ανθρώπινη κινητικότητα όσον αφορά την αλλογικότητα, ήταν πάντοτε σταθερή 2,9 με 3,3% του παγκόσμιου πληθυσμού κάπου εκεί κυμαίνεται σε πραγματικούς όρους θα είναι περισσότεροι άνθρωποι έτσι δηλαδή αυτό το 3% θα κινητοποιήσει και άλλους και δεν θα έχει κατανεμηθεί ομοιόμορφα. Με αυτή λοιπόν την κατάσταση θα πρέπει να ασχοληθούμε. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρξουν 7 εκατομμύρια Αφρικανοί που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Δεν το ξέρω. Πρέπει όμως να σας πω ότι αν αυτό ισχύει, αυτό θα είναι ένα ισχνό, ένα θα χλωμιάζει μάλλον στο ποσοστό που υποδέχτηκαν στο Λίβανο στην αρχή της Συριακής κρίσης. Δεν λέω ότι είναι καλό έτσι, αλλά η σύγκριση μεταξύ αυτού που συνέβη στο Λίβανο θα ήταν αν σαν ολόκληρος ο πληθυσμός του Καναδά πήγαινε μια νυχτή στις Ηνωμένε Πολιτείε. Και ακόμα και αυτό σαν αναλογία δεν φτάνει. Χρειαζόμαστε λοιπόν να έχουμε μια γενική εικόνα, μια σφαιρική εικόνα και να αναρωτηθούμε τι πρέπει να κάνουμε για να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Οπότε και πάλι ξαναλέω, δεν ξέρω αν θα έρθουν 7 εκατομμύρια Αφρικανοί στην Ευρώπη, αλλά αυτό που ξέρουμε για τη μετανάστευση είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία τη μετανάστευση είναι εσωτερική. Δηλαδή, ο κόσμο μετακινείται στο εσωτερικό τη χώρα του πρώτα, είναι επίση περιφερειακή στο Νότο το φαινόμενο της είναι επίσης τεράστιο και οι χώρες αυτές δεν είναι μόνο χώρες προέλευσης και αν συζητήσετε ας πούμε με Αφρικανούς ομολόγους θα ήταν πολύ χρήσιμο να μοιραστείτε μαζί τους ε, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζετε εσείς ως χώρα προορισμού γιατί έχουν και στο εσωτερικό τους παράνομους μετανάστες και αυτοί που είτε προσπαθούν να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης ή προσπαθούν να τακτοποιηθούν. Έχετε λοιπόν αρκετά κοινά αν παρακάμψετε στερεότυπα σε σχέση με τις χώρες προορισμού, προέλευσης, χώρες ε, διέλευσης κλπ. Η κινητικότητα λοιπόν είναι αρκετά κυκλική και αφορά όλους μας. Τώρα, υποχρεωτική ή όχι η εθελουσία εθελοντική αλληλεγγύη. Δεν ξέρω τι να σας πω εδώ. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι η Σύμβαση για την Μετανάστευση προβλέπει κάποιες εγγυήσεις. Δηλαδή ένα άτομο το οποίο διώκεται έχει βεβαίως κάθε δικαίωμα να διασχίσει τα σύνορα παράνομα. Έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει αν τη στιγμή που είναι διωκόμενος. Μπορεί να το κάνει νόμιμα, αλλά βέβαια εντάξει, πολλέ δεν τα καφένει καν χάνει τη ζωή του. Και η σύμβαση προβλέπει βεβαίως και κάποια κατανομή, κάποια κατανομή του βάρους ή του φόρτου. Γιατί, ξαναλέω οι Σύριοι που ήρθαν, δεν ήρθαν λόγω συνόρων, αλλά λόγω γεωγραφίας. Γιατί λοιπόν η του φορτου γιατι ξανα οι συριοι που ηρθαν δεν ηρθαν λογω συνορων αλλα λογω γεωγραφιας γιατι λοιπον η γεωγραφια θα έπρεπε να καθορίζει το ποιος έχει την ικανότητα ή τη δυνατότητα να διασώσει αυτούς που να αντιμετωπίζουν κάποια ανάγκη. Και είναι δυτή, είναι αφήσιμη, μάλλον δυτή η αλληλεγγύη. Αλλά και πάλι θα μιλήσω για την Ευρώπη, γιατί νομίζω ότι αυτά είναι θέματα τα οποία είναι εσωτερικά ίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχαμε και το βραβείο Νόμπελ που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο νομίζω το άξιζε. Τώρα βέβαια να πω ότι για αυτό το θέμα της μετανάστευσης, το οποίο αντιμετωπίζω εδώ και τρεις μήνες, περιλαμβάνει πολλά στοιχεία που αφορούν την καθημερινότητα Έχουμε θέματα υποδοχής και πολλά άλλα θέματα, αλλά όσον αφορά τι πολιτικές, αυτό που θα μπορούσα να πω και από νομική μάλιστα σκοπιά, ότι η υπεργολαβία όσον αφορά τις ευθύνες δεν είναι ένας αποδεκτός τρόπος απεμπόλησης ευθύνης. Η ευθύνη παραμένει. Έτσι, και δεν μπορώ να πω και κάτι παραπάνω. Και ταυτόχρονα να σας πω ότι την παραπάνω εβδομάδα θα πάω στη Ρώμη και ελπίζω εκεί να κατανοήσω κάπως καλύτερα το θέμα της θαλάσσιας ε, διάσωσης, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ακτές της Λιβύης. Γιατί τώρα δεν είμαι σε θέση βεβαίως να εκφράσω προσωπική άποψη για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Λουίζ. Λότι, θέλετε να κάνετε ένα σύντομο σχόλιο ίσως για τη Λιβύη. Θα βοηθούσε. Ένα από τα πλεονεκτήματα της εθνής μας ε, εκδήλωσης ήταν και το γεγονός ότι αναδείχθηκε ε, η ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής μας και της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Όμως η Μπάρμπαρα Σπινέλη έθεσε κάποια πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Θα ήταν καλό αν γίνεται να τα απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι νομίζω ότι η Αντιπρόεδρος ε, Μογκερίνη ασχολήθηκε με πολλά θέματα χθες στην παρέμβαση της και αφορούσαν όλα την ε, εξωτερική διάσταση της ε, ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Να απαντήσω σε ορισμένα από τα σχόλια που ακούστηκαν. Εμείς συμμετέχουμε στην περιοχή στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων γιατί αυτή είναι που καθιστά θύματα τους ανθρώπους, που πληρώνουν υψηλά ποσά και διακινδυνεύουν τη ζωή τους. Ε, ασχολούμαστε λοιπόν με τρόπους που μπορούμε να ε, σταματήσουμε τις ε, δραστηριότητες αυτών των ανθρώπων με μια σειρά από μέτρα. Συνεργασία με αρχές, ε, παροχή βοήθειας, συνδρομής, ε, εκπαίδευση, για να σπάσουμε αυτό τον κύκλο ε, και να εμποδίσουμε αυτά τα κυκλώματα του οργανωμένου εγκλήματος να εκμεταλλεύονται ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και αυτό το κάνουμε με όλους τους εταίρους μας, τη Λιβύη και άλλους. Ολιστική προσέγγιση, βεβαίως μια τέτοια προσέγγιση ακολουθούμε βλέπουμε τη μετανέστευση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στο, στην, και στη συγκεκριμένη περίπτωση μαζί με τους εταίρους μας από την ε, Αφρική. Τους αποκαλούμε μάλιστα αμοιβαίους κοινού στόχους και δεσμεύουν και εμάς αλλά και τους, τις τρίτες χώρες εταίρους μας. Και η εμπειρία που έχουμε συλλέξει στο πλαίσιο ε, της εταιρικής σχέσης που ε, συζητούμε πιο συχνά και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ενδεχομένω πιο πολύ, ε, αφορά ακριβώς ε, το να λαμβάνουμε υπόψη μα τι ιδέες, τι ανάγκες και των εταίρων μας. Και δεν μιλώ μόνο για χρήματα και κονδύλια, αλλά μιλώ για όλους τους τομείς πολιτικής στους οποίους μπορούμε να δώσουμε βοήθεια και όχι μόνο στη μετανάστευση, σε πολλούς τομείς πολιτικής. Και ένα από τα βασικά διδάγματα, ε, ε, ε αυτό είναι ένα από τα βασικά διδάγματα που ε, μεταφέραμε και στη Νέα Υόρκη. Τον, την ανάγκη να υπάρξει μια νέα, ένα νέο είδος εταιρικής σχέσης τόσο με τις αφρικανικές χώρες αλλά και όσο και με χώρες από άλλες περιφέρειες του πλανήτη. Να υπάρχει δηλαδή μια στάθμιση του τι ακριβώς ε, χρειάζεται. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τα ριζικά αίτια που βρίσκονται και στο επίκεντρο του, του προβλήματος. Είναι πολυδιάστατο και περίπλοκο το θέμα αυτό από τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων ε, σε, στις άλλες χώρες, τη, τη φτώχεια, την κλιματική αλλαγή, την ε, επιστημιστική ασφάλεια. Βεβαίω, λοιπόν, υπάρχει ανάγκη να λαμβάνονται βραχυπρόθεσμα μέτρα, όπω κάνουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χρειάζονται να λαμβάνονται και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Και για το σκοπό αυτό έχουμε συστήσει και αυτό το Trust Fund, προκειμένου να δίνεται βοήθεια σε χώρες εταίρους μας. Ε, προσπαθούμε να ε, εντάξουμε και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης το οποίο έχει ως στόχο να προσελκύσει ε, επενδυτές, ιδιωτικά κεφάλαια, προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Γιατί αυτό μας λένε οι χώρες εταίροι μας. Απασχόληση που θα οδηγήσει και σε μεγαλύτερη ασφάλεια. Άρα αυτό ε, δεν έρχεται σε αντίθεση, η δική μας προσέγγιση καθόλου δεν έρχεται σε αντίθεση με την προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί σε επίπεδο ΟΗΕ. Ε, και αυτό είναι το, το, το, το, το, γενικό σκεπτικό όλης της δράσης μας. Υπάρχει και η Σύνοδος ε, Κορυφής με την Αφρική φέτος. Βασικός στόχος είναι η αύξηση των θέσεων εργασίας. Πολλοί πάντοτε θα μετακινούνται, αλλά αυτό δεν είναι, δεν είναι το, το θέμα που μας απασχολεί. Βεβαίως κάποιοι μπορεί να θέλουν να φύγουν, άλλοι όμως και αυτοί που θέλουν να μείνουν στις αιστείες τους, στις πατρίδες τους, πρέπει να έχουν δουλειές, πρέπει να έχουν καλύτερες συνθήκες ε, διαβίωσης βιωτικού επίπεδου. Ε, αυτό αφορούν και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι που έχουμε θέσει. Όσον αφορά την επικοινωνική πολιτική, ε, πράγματι ε, χρειαζόμαστε μια καλύτερη, μια βασισμένη σε στοιχεία προσέγγιση. Πάντως, ακόμη και εκεί που υπάρχει μια τέτοια προσέγγιση, ακολουθείται μια τέτοια προσέγγιση, δεν, δεν, δεν αρκεί αυτό από μόνο του για να αλλάξουν οτροπίες αντιλήψεις των ανθρώπων. Για τη Λιβύη είναι, προφανώς, είναι προφανές ότι τα πράγματα είναι ρευστό, ρευστά. Ε, εκρεμεί μια πολιτική διευθέτηση του, ε, των προβλημάτων που υπάρχουν εκεί. Αυτό που προσπαθούμε πάντοτε εμείς να κάνουμε και με τη Σάφια είναι ε, να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές όπου και αν αυτές βρίσκονται. Ε, πάντως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκεται στο επίκεντρο των όσων κάνουμε. Και ε, η εκπαίδευση της ακτοφυλακής ε, αφορά 130 ε, ανθρώπους ακτοφύλακες. Αυτοί τα στελέχη της ακτοφυλακής περνούν ακριβώς μέσα από έναν κύκλο εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό δεν είναι αρνητικό. Αντιθέτω άνθρωποι που θα έχουν εκπαιδευτεί θα μπορούν και να παρακολουθούν ε, πώς και σε ποιες περιπτώσεις ε, ε, παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα. Κάποιοι μάλιστα αναφέρθηκαν στα 90 εκατομμύρια που έχουν ε, διατεθεί για αυτό το Trust Fund για την Λιβύη. Ο στόχο στόχος είναι να βελτιώσουμε τους, τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων στα κέντρα όπου βρίσκονται. Ε, μέτρα υγιεινής, τρόφιμα, ε, κουβέρτες, ε, ρουχισμό, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εκεί κατευθυνούν τα χρήματα αυτά. Αφετέρου, ε, στόχος μας είναι αφού οι άνθρωποι διασωθούν και επιστραφούν στη Λιβύη θα έχουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας στη Λιβύη και με, χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι δεν θα, δεν και ε, περαιτέρω δράσεις. Ε, αυτό που μας απασχολεί είναι πάντοτε να ε, γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σόφη και Μπάρμπαρα, θέλετε να επανέλθετε, ε, να ξαναπαρέμβετε. Φαντάζομαι ότι είναι για, για τη Λιβύη. Ναι. Αυτό που λέτε έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την παρουσίαση που παρακολουθήσαμε πριν από μερικέ ε, εβδομάδε από του γιατρού χωρί σύνορα, που είναι η μόνη οργάνωση που βρίσκεται επί τόπου. Η εικόνα που μα περιέγραψαν λοιπόν ήταν τελώ διαφορετική από, από αυτή που μα περιγράφετε εσεί. Μα περιέγραψαν μια κόλαση. Και μα είπαν ότι μα δόθηκαν 90 εκατομμύρια ευρώ. Πέραν το ότι έχω πολλές αμφιβολίες για το κατά πόσο η ακτοφυλακή της Λιβύης μπορεί να ε, αποτελέσει το κέντρο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, το βασικό ερώτημα είναι... Ε, ας το πούμε για, την, για την ε, διευκόλυνση συζήτηση. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε αυτά τα 90 εκατομμύρια ευρώ για να, για να τους ε, στεγάσουμε και να τους εντάξουμε εδώ στην Ευρώπη ή γιατί δεν τους δεν δίνονται αυτά τα χρήματα τουλάχιστον για να επιστραφούν στις πατρίδες τους και δίνονται για να εγκλωβιστούν στην ε, Λιβύη. Πάρμπαρα πολύ γρήγορα, για να απαντήσει η Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη από την, απόφαση, από την απάντηση εκπροσώπου της Κομισιόν. Και θέλω να αναφέρω αυτό που είπε ο κύριος Κόμπλερ για την κατάρτιση των ε, ακτοφυλάκων. Εγώ ε, δεν συνιστώ να συνεχιστεί αυτή η ακτοφυλακή, η ε, κατάρτιση των Λίβιων ε, ακτοφυλάκων. Θα πρέπει στην επιχείρηση Σοφία να συμμετάσχει και ο ΙΕ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μετά την κατάρτιση όλα θα είναι τέλεια. Αν πάτε στη Λιβύη θα δείτε Λίβιους ε, ακτοφύλακες που σπρώχνουν τους, άνθρες, τους ανθρώπους στη θάλασσα για να πνιγούν. Μπορείτε να το γκουγκλάρετε στο YouTube. Μερικοί μάλιστα ε, τους ε, πυροβολούν κιόλα. έτσι. Άρα δεν είμαι σε καμία περίπτωση ικανοποιημένη με την απάντησή σας. Λότι. Και οι δύο μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα. Ζητάω από τους δύο συναδέλφους να απαντήσουν. Ε, δεν έχουμε τακτικές επαφές με την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ε, αυτό είναι το πρόβλημα και θα ήθελα να ακούσουμε μια απάντηση τώρα. Το ακούω συνέχεια αυτό από του ευρωβουλευτέ, να παραπονιούνται κτλ. Είτε ο κ. Αμπρόζη είτε η Λότη. Κάποιο από του δύο να απαντήσει. Σύντομα. Εμείς ε, είμαστε σε επαφή με την ε, Λιβύη. Ποτέ δεν φύγαμε από τη Λιβύη. καθημερινά λειτουργούμε στα κέντρα κράτησης. Ξέρουμε πολύ καλά περί πρόκειται. Ας μιλήσουμε ανοιχτά και ειλικρινά. Καταρχάς, καθημερινά στη Λιβύη αντιμετωπίζουμε μία δέσμη αδύνατων επιλογών. Όλες είναι αδύνατες. Αν έπρεπε εγώ να επιλέξω κάτι, αν μιλούσαμε για την δική μου τη χώρα, την Ιταλία, δεν θα επέλεγα τίποτα από όλα αυτά. Αλλά το, δεν μιλάμε για την Ιταλία, μιλάμε για τη Λιβύη. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Καθημερινά παλεύουμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε ποια είναι η λιγότερο καταστροφική ή επιβλαβής απόφαση που μπορούμε να πάρουμε. Δεύτερο. Και εμείς δεν καταρτίζουμε την, τους ακτοφύλακες, δεν είμαστε αυτοί. Δεν έχουμε καμία σχέση με την για την κατάρτιση, έτσι. Κάνουμε κάποια κατάρτιση για τις πρώτες βοήθειες και την ε, διάσωση στη θάλασσα που παρέχουν στους ανθρώπους στα σημεία αποβίβασης. Έτσι, τίποτα άλλο. Αλλά πριν από δύο ή τρεις εβδομάδες, η μισή Ευρώπη, η πολιτική πολιτικη αρχικη οι εφημερίδες παραπονιόνταν για τις ΜΚΟ που διασώζουν μετανάστες από την ακτή της Λιβύης. μας αποκαλούσαν τα ταξί της Μεσογείου που βοηθάμε τους διακινητές και που μας πληρώνουν οι διακινητές. Ακόμα και την ε, μη κυβερνητική οργάνωση που αναφέρατε, έτσι, που βοηθάει τα παιδιά κτλ. Έχουμε επίσης ε, πολύ μεγάλες επιφυλάξεις ε, για την Λιβική Ακτοφυλακή που κάνει επιχειρήσεις έρευνα και διάσωση. Επομένω, το ερώτημά μα είναι τι να κάνουμε, ποια είναι η εναλλακτική. Είμαστε, α πούμε, τα ταξί τη Μεσογείου που υποστηρίζουν του διακινητέ, Η λιβική ακτοφυλακή είναι προβληματική. Δεν τελείωσα, περιμένετε, ακούστε με. Τι να κάνουμε λοιπόν εμεί τι κάνουμε. Πώ αποφεύγουμε το θάνατο των μεταναστών στα νερά τη Λιβύης. Γιατί αν κανένα δεν κάνει τίποτα εκεί πέρα, ο κόσμο θα πεθάνει. Επομένως, η επιλογή που κάναμε μπορεί να αφισβητήσετε, είναι οριακή. Τέλο πάντων, με αυτά τα δεδομένα, το καλύτερο που κάνουμε είναι αυτό που θα σας πω. Είναι μειώνουμε όσο μπορούμε ε, τα βάσανα των ανθρώπων αυτή τη στιγμή τους ε, διασώσουμε. Ε, ναι, υπάρχουν πολλοί θάνατοι βέβαια, αλλά υπάρχουν και 60.000 άνθρωποι που διασώζονται και που δεν τους πετάμε πίσω στη θάλασσα. Έτσι. Προσπαθούμε να μειώσουμε τα βάσανα αυτών των ανθρώπων προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε και στα κέντρα κράτησης που εμείς ως ΟΗΕ και ως ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, δεν τα θέλουμε, δεν τα υποστηρίζουμε αυτά τα κέντρα κράτησης. Αλλά με βάση την ε, νομοθεσία της Λιβύης προβλέπονται κέντρα κράτησης για τους λαθομετανάστες. Δεν μας αρέσουν, αλλά έτσι είναι. Η ποινικοποίηση των ε, λαθρομεταναστών είναι μάλιστα και μια νομική αρχή που χρησιμοποιείται και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι. Ε, χρησιμοποιούν ε, ευρέω τις ευρωπαϊκές χώρες την κράτηση για τους λαθρομετανάστες. Φυσικά εμείς είμαστε κατά, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να μειώσουμε τα προβλήματα των ανθρώπων στα κέντρα αυτά. Και τέλος και τελευταίο. Δεν υπάρχει επιστροφή από την Ευρώπη στη Λιβύη. Αυτοί, αυτοί οι άνθρωποι διασώζονται στα ύδατα της Λιβύης. Είναι ακόμα στην επικράτεια της Λιβύης. Υπάρχει όμως που υπάρχουν πολλές θελοντικές επιστροφές από τα κέντρα κράτη της Λιβύης και από τα υπόλοιπα σημεία της Λιβύης που πάνε σε εμάς είτε στον ΟΗΕ και λένε «Κοιτάξτε, θέλουμε να φύγουμε τη Λιβύη, θέλουμε να επιστρέψουμε στην πατρίδα μας». Είναι τέλεια η κατάσταση. Όχι. Αλλά η Λιβύη δεν είναι μια, ένας παράδεισος, μια ιδανική κατάσταση. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Εγώ αντιδρούσα στις ε, δηλώσεις της κυρίας ε, Λότη ε, από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Καταλαβαίνω αυτά που λέτε, αλλά εγώ απευθυνόμουν στην κυρία Κρούτσεν και μέσω αυτής στις 28 κυβερνήσεις των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Καταλαβαίνω αυτά που λέτε εσείς. Εσείς αντιμετωπίζετε τις συνέπειες όπως μπορείτε. Εγώ μιλάω και απευθύνομαι στους πολιτικά υπεύθυνους, την Κομισιόν, την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, εσείς φυσικά δεν είσαστε πλήρως υπεύθυνος για αυτές τις αποφάσεις. Είστε σε κάποιο βαθμό. Είσαστε συνένοχος σε κάποιο βαθμό. Και όταν μου λέτε, ναι, είναι προβληματική η κατάσταση λιγάκι, αλλά την αντιμετωπίσουμε και καταρτίζουμε τους ακτοφυλακές, ε, με ενοχλεί λιγάκι. Και ο κ. Αμπρόζη επιβεβαιώνει ότι η κατάσταση είναι άθλια. Δεν υπάρχουν καλές επιλογές καθόλου. Υπάρχουν αυτές οι διαφορές λοιπόν ανάμεσα σε αυτές τις κουβέντες περί υποδοχής στην ε, περιοχή και ότι είναι θαυμάσια αυτή η λύση και στην πραγματικότητα και τις εικόνες από την πραγματικότητα που βλέπουμε. Υπάρχει μια άβυσος μεταξύ τους. Δεν μπορώ και τα δύο είναι αλήθεια. Σόφι, συνάδελφοι, Μπάρμπαρα, όλοι σας είναι το άθλιο καθήκον μου για ένα τόσο ε, σημαντικό θέμα ειδικά. Ε, σας έδωσα βεβαίως το λόγο γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα ε, και η Λότη είναι σημαντικό να απαντήσει και ευχαριστώ τη Λότη για τη συνεισφορά της, αλλά έτσι προέκυψε σε αυτή τη φάση, αλλά το πρόβλημα είναι το εξής. δεν μπορούμε να αφιερώσουμε συζήτηση στο θέμα τη έρευνα και διάσωση. Θα το κάνουμε στι 12 του μηνό και θα προσκαλέσουμε του πάντε. Σα παρακαλώ και εκεί τότε θα επικεντρωθούμε στην διάσωση. Σήμερα καλέσαμε τη Λουίς Άρμπορ για να μα μιλήσει για όλο τον κόσμο, για το θέμα το σημερινό. Ε, αν ε, επικεντρωθούμε αποκλειστικά στη Λιβύη, δεν είναι σωστό, δεν είναι δίκαιο. Θα ήθελα να τελειώσουμε αυτό το σημείο. Πρέπει να το είχαμε τελειώσει μάλιστα πριν από 15 λεπτά. Νομίζω όμω ότι σεβάστηκα τις ανάγκες όλων. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όμως άλλο. Στις 12 Ιουλίου θα έχουμε το θέμα της έρευνας και διάσωσης και θα μιλήσουμε για τη Λιβύη ενδελεχώς. Ε, θα είναι και η Λουίζ Άρμπορ. Ελπίζω όλοι σας να είστε. Τότε μπορούμε να συζητήσουμε ενδελεχώς αυτά τα θέματα. Θα τσεκάρω πάλι το πρόγραμμα γιατί θέλω να είμαι σίγουρος ότι θα έχετε όλο τον χρόνο για να μιλήσετε για αυτά τα θέματα. Και θα το επιβεβαιώσω μέσω των συντονιστών σήμερα. Λουίζ. Η Λουίζ κανονικά πρέπει να έχει φύγει. Την ανάγκασα να παραμείνει για να της πω πόσο την ευχαριστώ για τη συνεισφορά της. Ε, εμπλεκόμαστε επίσημα στη διαδικασία της Νέας Υόρκης. Θα τα διαβάσω τώρα όλα αυτά. Θα πάτε και στο Μεξικό, από ό,τι ξέρω, και οι εμπειρογνώμονες από την άλλη οργάνωση θα πάνε εκεί και άλλες ε, αντιπροσωπείες επίσης και από τις άλλες ε, επιτροπές. Θα τα πούμε εκεί. Ευχαριστώ, Λουίς, για τη συνεισφορά σου. Ευχαριστώ επίσης και τη Λότη από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τον συνάδελφο Αμπρόζη. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση, συνάδελφοι, για τη Λιβύη, ειδικά στις 12 Ιουλίου. Μπορούμε να ξανασυζητήσουμε το πρόγραμμα εκείνης της ημέρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ στην και για το ενδιαφέρον σας. <laughs> colleagues, I know this is very tight and people are... Um, we have a short meeting and I know people have to Δεν έχουμε χρόνο. Ξέρω θα πρέπει να πάτε και στα σπίτια σας. Οπότε πάμε στο επόμενο σημείο, στο σημείο 10. Παρουσίαση μιας μελέτης της Νοτάσια Ζάουν και Βιολέτα Μορέ, ε, Μορένο Λάξ μελέτη που ζητήσατε εσείς οι συντονιστές για την εφαρμογή των αποφάσεων Συμβουλίου του 2015 για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας. Είναι προφανές περί τίνος πρόκειται και του ουρού θα πάω σε δύο, στις δύο, δύο Έχουν διαφάνειες Παρακαλώ, έχετε λόγο. Ωραία, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την Επιτροπή σας για την υποδοχή. Με χαρά βρισκόμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα της μελέτης επανακατάστασης στην Επιτροπή σας. Πριν να αναφέρουμε στοιχεία για τα σχέδια μετακατάστασης, να σας μιλήσω για τα κυριότερα σημεία. Έχουμε τρεις σημαντικές αποφάσεις, δύο υιοθετήθηκαν μετά το καλοκαίρι του 2015, μία απόφαση το 2016, που, προσαρμο, που προσέρμοσε δύο προηγούμενες στο νέο πλαίσιο της συμφωνίας με την Τουρκία. Είχαμε αυτές αποφάσεις λοιπόν για να ελαφρύνουμε την πίεση στην ε, Ιταλία και την Ελλάδα. Έχουμε τρεις μήνες για να υλοποιήσουμε το 90% του αρχικού έργου τη στιγμή που έχουμε μόνο 10% με καταστάσεων που έχουν υλοποιηθεί. Αυτό αφορά όλε τι χώρε μέλη, εκτό Δανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, Λιχτεστάιν, Νορβηγία, Ελβετία κλπ. Διαχειριζόμαστε τις ποσοστώσεις αναχώρα και μια κλίδα κατανομή, κατανομής λαμβάνοντας υπόψη δύο στοιχεία, ΑΕΠ και συνολικό πληθυσμό, όπως επίσης ποσοστό ανεργίας και δυνατότητα υποδοχής. Είχαμε δυσκολίες και νομικές, αλλά και υπό την αρχή της μη διάκρισης για τους πρόσφυγες όσον αφορά την υποδοχή και την πρακτική της εφαρμογή, επειδή ήταν δύσκολο να προκαταβάλουμε ποιες εθνικότητες είχαν δικαίωμα να μετεγκατασταθούν τους επόμενους μήνες. Η κατανομή των ποσοστώσεων μεταξύ των χωρών ήταν ανισοβαρή, θα μας πει περισσότερα η Νατάσα. Ξεκίνησε η διαδικασία παραβίασης ε, η Κομισιόν κατά Ουγγαρίας και Τσεχίας την περσμένη εβδομάδα, οι οποίες, χώρες οι οποίες αντιτάχθηκαν ή ήταν διστεκτικές στην εφαρμογή των αποφασισμένων. Νατάσα, η ηταν δυστεκτικες στην εφαρμογη των αποφασισμενων νατασα η επομενη Α δούμε τις χώρες που τα εφάρμοσαν αυτά σωστά και τις χώρες που δεν τα πήγαν και τόσο καλά. Η Μάλτα είναι η μοναδική χώρα που μέχρι τώρα εκπλήρωσε το καθήκον τη. 100% μετακαταστάσεων. Αλλά οι υπόλοιπε χώρες όχι. Οι συνδεδεμένε χώρες και αυτές τα πήγαν καλά. Φινλανδία, Ιρλανδία επίσης τα πήγαν καλά και άλλε χώρε καλούτσικα τα πάνε, αλλά εντάξει. Όχι θαυμάσια. Επόμενη διαφάνεια. Χώρες μέλη που δεν τα πήγαν και τόσο καλά. Βλέπουμε ότι δεν έχουν κάνει καμιά μετεγκατάσταση κάποιες χώρες. Αυστρία, Ουγγαρία, Πολωνία και Τσεχία είναι σχεδόν στο 0. 0% δηλαδή των ε, ποσοστώσεων τους. Κάποιες άλλες χώρες η Σουηδία ας πούμε, τα πάει σχετικά καλά. Αλλά Σουηδία και Αυστρία είχαν κάποιες παρεκκλήσεις για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό εξηγεί το ότι δεν τα πήγαν και τόσο καλά. Αλλά βέβαια δεν εξηγεί το μηδενικό ποσοστό της Αυστρίας. Επόμενη διαφάνεια. Συλλέξαμε κάποια δεδομένα κάναμε συνεντεύξεις, είχαμε επαφές με τα Εθνικά Σημεία Επαφής, ΜΚΟ, χώρες μέλη και είδαμε ότι καταρχάς η πολιτική στήριξη είναι πολύ σημαντική ώστε να λειτουργήσει η μετακατάσταση και όπως είπαμε ήδη, οι χώρες του Βίζεγκρατ εξ αρχής ήταν κατά αυτής της απόφασης και δεν πήγαν και πολύ καλά στην εφαρμογή της απόφασης. Επειδή δεν υπήρχε πολιτική στήριξη οι χώρες μέλη που το αποδέχτηκαν τα πήγαν καλά, το οποίο μας καταδεικνύει και μας αποδεικνύει ότι η πολιτική βούληση, η πολιτική στήριξη είναι απαραίτητη. με τα δυνατότητα αποδοχής Το 2015 κάποιες ε, χώρες δέχτηκαν κάποιες ή αρκετές αιτήσει, αλλά είχαν κάποια προβλήματα όσον αφορά την υποδοχή. Και υπάρχει κάποια συγκεκριμένη δυναμική εδώ, γιατί υπάρχουν χώρες όπως η αρκετες αιτησει αλλα ειχαν καποια προβληματα οσον αφορα την υποδοχη και υπαρχει καποια συγκεκριμενη δυναμικη εδω γιατι υπαρχουν χωρες οπως η φιλανδια που δέχτηκαν πολλές αιτήσει το 2015, και είχαν σημαντική αύξηση και βρισκόταν στη δικασία επεξεργασία, που έγινε όμω που ολοκληρώθηκε τόσο γρήγορα που πλήρωσαν, που κατάφεραν να συμπληρώσουν το, τις ποσοστώσεις τους για μετακατάσταση. Έχουμε επίσης και τους πιο ευάλωτους και τις αντίστοιχες αιτήσει, ασυνόδευτα παιδιά κτλ. Υπήρχαν χώρες που είπαν δεν είχαν επαρκή δυνατότητα υποδοχής Έχουμε επίσης και τις αντιλήψεις σε σχέση με τις απειλέ όσον αφορά την ασφάλεια, κάτι το οποίο οδήγησε επίσης σε χαμηλότερη μετεγκατάσταση. Και οδήγησε κάποιε χώρε να εξαιρέσουν κάποιους ετώντε. Και αυτό ήταν πολύ προβληματικό γιατί δεν ανέφεραν για ποιους λόγους ε, απέκλειναν συγκεκριμένου ετώντε να εξηγήσω τα προβλήματα στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Υπάρχουν βέβαια κάποιες εξωτερικές προκλήσεις. Υπάρχει καθυστέρηση όσον αφορά τι μεταφορέ, υπάρχουν ατεκμηριώτε απορρίψει, υπάρχει ελλειπή τεκμηρίωση. Υπάρχουν επίση περίπλοκε τοπικέ διαδικασίε, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Είχαμε ένα πρόβλημα υπερσυγκέντρωση, όπου οι ετώντε στα νησιά δεν είχαν πληροφόρηση για την διαδικασία. Στην Ιταλία είχαμε πρόβλημα με την μετεγκατάσταση και τι τοποθεσίε, όπου πήγαιναν οι πρόσφυγε σε διαφορετικέ περιφέρειε, ανάλογα με την κατάσταση πρόοδου τη αίτησή του. Αυτό τους πρόσφυγες να μην έχουν αρκετές πληροφορίες για την κατάσταση της αιτησής τους, για το που θα πάνε και κάποιες πληροφορίες που λάβαναν ήταν μόνο από τη Wikipedia σε σχέση με, το, με την τοποθεσία με την κατάσταση. Και δεν είχαν δυνατότητα νομικής βοήθειας. Δεν λάμβαναν καμία πληροφορία δηλαδή σχετικά. Ούτε καν ήξεραν σε κάποιε περιπτώσει σε ποια χώρα θα πήγαιναν. Thanks. Εκτός από το σύστημα μετακατάστασης, ε, εξετάσαμε και αυτή την προσέγγιση με τα hot spot που είχε ανακύψει ad hoc βεβαίως όταν προέκυψε η κρίση. Ε, πρώτον, πρώτος στόχος λοιπόν ήταν η ταυτοποίηση των υποψηφίων προς μετεγκατάσταση. Από την υπογραφή όμως της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας ε, τα hot spot ε, ε, ειδικεύονται στον έλεγχο της μετανάστασης. Ε, σε αυτό το πλαίσιο ε, η Frontex έχει πολύ πιο ηγετικό ρόλο σε σχέση με την ΙΑΣΟ που θα έπρεπε κανονικά να είναι ο οργανισμός που θα είχε τεθεί επικεφαλής. Στην πραγματικότητα είναι πλέον ε, ο, η, το, νέο καθεστώς ε, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή ε, είναι ο μόνος κανονισμός που ορίζει ποιες είναι, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των Εθνικών Ομάδων Διαχείρισης Μετανάστευσης και ως προς τη λογοδοσία. Σημαντικότερος είναι ο ρόλος της Frontex Άλλοι οργανισμοί βεβαίω παρεμβαίνουν και εκείνοι στα hotspot και έχουν ε, συγκεκριμένες επιπτώσεις στο τι γίνεται στα hotspot. Eurojust, Europol, καταπολέμηση οργανωμένου εγκλήματος, ε, λήψη αποφάσεων ε, μετεγκατάστασης. Πολλές φορές όμως υπερβαίνουν τους, ε, η Frontex υπερβαίνει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του και το έχει πει αυτό και ο Ευρωπαίος Δημοσιολαβητής. Το γεγονό ότι δεν υπάρχει λοιπόν ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο είναι ένα πραγματικό μειονέκτημα ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν ούτε μηχανισμοί παρακολούθησης ούτε προσφυγή, χρήση προσφυγής, σε ένδικα μέσα ε, και έτσι έχουν ε, υπάρξει ε, παραβιάσεις που έχουν παρατηρήσει πολλοί παρατηρητές και η δική σας επιτροπή. Υπάρχει λοιπόν μια συνύπαρξη των hot spot και της μετακατάσταση με τις μεταφορές Δουβλίνου. Στην Ιταλία για παράδειγμα ο αριθμός των, των ανθρώπων που περνάνε μέσα από τα hot spot είναι μεγαλύτερος από ότι στο, σύστημα του, του Δουβλίνου. Τα λέω λίγο γρήγορα για να μην καταχαστώ το χρόνο σας. Ε, το σύστημα λοιπόν ε, έχει ως στόχο να ε, ε, επιτευχθεί μια καλύτερη διαχείριση και σε πολιτικό επίπεδο της μεταναστευτικής κρίσης. Αποτελεί ένα, μια πρώτη προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την, τον επιμερισμό των ευθυνών ε, σε συμφωνία και με, την, με το άρθρο 80 της Συνθήκης για, την, για, για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την σχετική αλληλεγγύη που ε, προβλέπεται. Τα βασικά ε, αρνητικά όμως πρέπει πρώτον να διορθωθούν προκειμένου το σύστημα αυτό να ε, ανταποκρίνεται στα θεμελιώδη δικαιώματα και στις ε, προβλέψεις της συνθήκης της Λισαβόνας για τη λειτουργία, και για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βασικά μειονεκτήματα που έχουμε εντοπίσει, θα σας πω πέντε, είναι πρώτον η απουσία πλήρους συμμετοχής των κρατών μελών. Κάτι που μετουσιώνεται σε απορρίψεις, σε υπερβολικούς ελέγχους, σε χαμηλό ρυθμό μεταφορών, όπως αναφέραμε ήδη. Κάτι που επιβραδύνει και ε, ε, υπονομεύει και την αποτελεσματικότητα ολόκληρου του συστήματος. Νομίζω ότι η, επιβράβευση της καλής πρακτικής αλλά και ε, η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης του συστήματος πρέπει να ενισχυθούν. Ε, κάτι που ε, θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό σε σχέση με τη διαδικασία που παραβάσει. Καλύτερα να δημιουργούνταν λοιπόν ένα σύνολο κινήτρων. Δεύτερον, τα δικαιώματα των ε, ε προσφύγων πρέπει να τεθούν, πρέπει να, είναι ανώτερα από οποιοδήποτε σύστημα, οποιοδήποτε κανονισμό του Δουβλίνου. Επίσης, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι ίδιοι προσφέρει θα εμπιστεύονται το σύστημα. Και ο εξορθολογισμός του, του εργαλείου αντιστοίχηση της ΕΑΖΟ είναι ένα πολύ καλό ε, εργαλείο που θα πρέπει να ενισχυθεί. Επίσης, ο ορισμός ε, καθηκόντων υποχρεώσεων όλων των ε, εμπλεκόμενων φορέων. Πρέπει αυτό να εξασφαλιστεί προκειμένου να ε, αποφευχθεί η υπερβολική, ο υπερβολικά γραφειοκρατικός χαρακτήρας των διαδικασιών. Αντί λοιπόν κάθε οργανισμός μόνος του, θα ήταν καλύτερο να υπάρχει ένας κανονισμός ο οποίος θα περιέγραφε τη διαδικασία στο σύνολό τη. Επίσης, πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το πρωτογενές δίκαιο, ιδίω με την ε, ε, χάρτα για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία να ελέγχονται ως προς την εφαρμογή τους. Και τέλος, το σημαντικότερο στοιχείο για, την, ε, για να γίνει θεσμική κατοχήρωση ενός συστήματος ε, με ε, ε, σε αντίθεση με αυτά που προβλέπει ο, ο κανονισμός του Δουβλίνου θα πρέπει να υπάρχει ε, ένας μηχανισμός, μόνιμος μηχανισμός κατάσταση προσφύγων. Αντί λοιπόν να ερχόμαστε και να, να ανταποκρινόμαστε σε κρίσεις υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να κατοχυρωθεί ένας μηχανισμός για το πώς θα κατανόημονται αυτού του είδους οι ευθύνε και τα βάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Κατευθείαν ε, ο εισηγητής, μάλλον θα δώσω λόγο στους αδέλφους, ο εισηγητής δεν είναι εδώ. Αλλά οποιοδήποτε συνάδελφος θέλει να κάνει ερωτήσεις ε, επί της έκθεσης, παρακαλώ, η Μπάρμπαρα. Ευχαριστώ πολύ την καθηγήτρια Λάξ, που τα ξέρει αυτά απ' έξω και Κάθε κείμενο που γράφει, για μένα είναι σημείο αναφοράς. Και εδώ μας παρουσίασε ακόμα μία μελέτη πολύ ενδιαφέρουσα. Αυτό το θέμα των μεταφορών του Δουβλίνου οι επιστροφές, ας πούμε, στην Ιταλία είναι διπλάσιες ή τριπλάσιες από τις μετεγκαταστάσεις. Επιστροφές από την Ιταλία, μάλλον. Να σας ρωτήσω το εξή για αυτό το θέμα. Υπήρξαν δικαστικές αποφάσεις και για την Ιταλία και για την Ελλάδα, όπου ζητούσαμε, ζητούσαν να μην μεταφερθούν μετανάστες και πρόσφυγες βάσει του Δουβλίνου στις χώρες τους, γιατί οι χώρες αυτές δεν ήταν στο ύψος που θα έπρεπε. Μία αφελής ερώτηση, μία ερώτηση αδαούς. Πώς αγνοήσαμε αυτές τις αποφάσεις του δικαστηρίου, πώς είναι δυνατόν. Και δεύτερον, και ένα άλλο σημείο που αναφέρεται στη μελέτη. που είναι η οικογενειακή επανένωση, που είναι μια προτεραιότητα. Προτεραιότητα σε σχέση, στα πλαίσια της μετεγκατάστασης. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να κάνουμε πάρα αυτά είναι πάντα η οικογενειακή επανένωση. Το επιβάλλει και το σύστημα του Δουβλίνου. Πρόσφατα υπήρξε μια συμφωνία μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας, μεταξύ των δύο κυβερνήσεων δηλαδή, των δύο χωρών αυτών, βάσει των, της, της οποίας συμφωνίας χιλιάδες πρόσφυγες που είχαν ήδη πάρει το καθεστώς που επέτρεπε την οικογενειακή επανένωση, δεν μπορούν να επανενωθούν με τις οικογένειές τους στη Γερμανία. Αν μπορέσουν να το κάνουν θα πρέπει να περάσουν πρώτα από μια πολύ επαχθή και πολύ α, μακρά διαδικασία. Κι όμως αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα που είναι η οικογενειακή επανένωση, πώς είναι δυνατόν πώς μπορούμε να το επιβάλλουμε. Το επιβάλλει ο νόμος. Και όμως για πολιτικούς λόγους συχνά το παραβλέπουμε, το αγνοούμε. Φαντάζομαι ότι η Γερμανία για πολιτικούς λόγους, προεκλογικούς λόγους. για αυτό το λόγο η Γερμανία επέβαλε στην Ελλάδα και η Ελλάδα δέχτηκε αυτή τη μείωση των ροών για λόγους οικογενειακής επανένωσης. Θα έπρεπε αυτές οι ροές να λάβουν χώρα δια νόμου. Ο νόμος το προβλέπει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μπάρμπαρα. Κυρία Βεργιά. Και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για αυτή τη μελέτη. Διερωτώ με, αν κάνετε τη μελέτη αυτή από νομικής πλευράς ή αν πήγατε επί τόπου για να κάνετε κάποιες διαπιστώσεις. Έχω τρεις ερωτήσεις. Εσείς στην έκθεσή σας ε, εστιάζεστε στους ευπαθείς πληθυσμούς και στη δυσκολία που μοιάζουν να, έχουν τα κράτη μόλι για να υποδεχθούν αυτούς τους ευπαθείς ανθρώπους. Ε, με βάση τις δικές μου πληροφορίες, στην Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, τα άτομα τα οποία σήμερα κρατώνται, βρίσκονται στα νησιά, είναι όλο και περισσότερο τέτοια ευπαθή άτομα. Συμφωνείτε με αυτή τη διαπίστωση? Και αν ναι, πώς μπορούμε να δράσουμε, ώστε να λάβουν αυτό το δικαίωμα στην προστασία. Δεδομένη της πορείας τους, νομίζω ότι είναι λογικό οι ενδιαφερόμενοι να αναγνωριστεί ότι υποφέρουν και ψυχολογικά. Υποτίθεται ότι ετοιμάζεται μια συμφωνία για να επιτρέψει την επιστροφή και αυτών των ατόμων, παρότι είναι ευπαθείς ενώ μέχρι τώρα προστατευόταν από το ευρωπαϊκό δίκαιο και από το διεθνές δίκαιο. Επίσης μιλήσατε για τις, τα ένδικα μέσα. Αν έχω σωστέ πληροφορίε, μοιάζει ότι δίνουμε όλο και περισσότερο την επιλογή, αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, στα άτομα αυτά, μεταξύ της δυνατότητας να υποφεληθούν από την εθελοντική επιστροφή ή να παρεντηθούν σε όποια ε, παραιτηθούν από το δικαίωμα της ε, προσφυγής και των ενδικών μέσων. Μου το επιβεβαιώνετε, συμβαίνει κάτι τέτοιο και επίσης, τέλος, υπάρχει μία συμφωνία που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ετοίμασε μάλλον ε, το Δεκέμβριο, συμφωνία με την Ελλάδα, όπου πιέζει την Ελλάδα σε ένα αντιφατικό σχήμα από ό,τι άκουσα. Από αυτά άκουσα. Από αυτά που άκουσα ε, χθε στην Ολομέλεια από τον Έλληνα Υπουργό Εσωτερικών. Εσείς ακούσατε για αυτό το σχέδιο δράσης που ετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα. Και αν ναι, τι επιπτώσεις θα έχει στα δικαιώματα των ενδιαφερομένων. Κατερίνα Κινίτσι. Αλλά θα είναι η τελευταία ερώτηση αυτή, γιατί έχουμε και ένα τελευταίο σημείο για τους ε, καταγγέλλοντες καταγγέλλοντε τη λειτουργία κτλ. Κατερίνα, τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Βιολένα Μορέτο Λάξ, την καθηγήτρια, για την ενδιαφέρουσα αυτή μελέτη. Είμαι Ιταλίδα. Ε, αισθάνομαι και εγώ ότι εμπλέκομαι σε αυτόν τον προβληματισμό και για τη χώρα μου υπάρχουν τις λειτουργίες Νομίζω ότι αναγνωρίζεται τώρα σε όλα τα επίπεδα ότι έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια για να υποδεχτούμε την τεράστια, τον τεράστιο βαθμό, τον τεράστιο αριθμό μεταναστών που φτάνουν στις ακτές μου, στις ακτές μας, της ε, Σικελίας κυρίως, γιατί είμαι Σικελία, έτσι. Φυσικά υπάρχουν λειτουργίε, φυσικά υπάρχουν ε, καθυστερήσει στην ε, διεκπαιρέωση των αιτήσεων ασύλου, αλλά η Ιταλία έκανε πραγματικά πολλά κυρίως για εκείνη την ε, κατηγορία ευπαθών που, ατόμων που είναι οι ανήλικοι, κυρίως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Πολύ σύντομα λοιπόν το ερώτημά μου είναι το εξή. Αναφερθήκατε πολύ σωστά στην μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου. Την περιμένουμε αυτή την μεταρρύθμιση όλοι μας. Αλλά παρόλα αυτά, με στάνομαι μηχανή απέναντι σε αυτή τη μεταρρύθμιση που ετοιμάζεται. Εσείς λέτε ότι έτσι όπως ετοιμάζεται αυτή η μεταρρύθμιση μπορεί να συνεισφέρει και να στηρίξει αυτές τις δύο χώρες, την Ιταλία και την Ελλάδα που κάνουν τη μεγαλύτερη προσπάθεια υποδοχής των μεταναστών. Εγώ, επαναλαμβάνω, έχω κάποιες αμφιβολίε και ερωτηματικά. Και κυρίως αναφέρομαι στους ανήλικους και του ασυνόδευτους ανήλικους. Κατά την άποψή μου, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι θα πρέπει να έχουν σε ό,τι αφορά ε, την κατάσταση οικογενική, επανε... οικογενική επανένωση και την αίτηση ασύλου, θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Ποια είναι η άποψή σα, λαμβάνοντα υπόψη και τη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου. Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Κυρία Μαρίνο Λάξ, θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Για την ερώτηση της κυρίας Σπινέλη, οι μεταφορές δουλειών που ξεπερνούν τον αριθμό μετεγκαταστάσεων. Είχαμε δύο υποθέσεις, δικαστικές στα Ρακέλ που αφορούσαν την Ιταλία και την Ελλάδα. Αν ερμηνευτούν σωστά και εφαρμοστούν σωστά, τότε οδηγούν βεβαίω στην de jure διακοπή του συστήματο μεταφορών του Δουβλίνου. Τουλάχιστον όσον αφορά τι μετε... τις, ε, οικογενειακέ επανενώσει και, τους... και τα συνόδευτα. Όπω μα έλεγε η Νατάσα προηγουμένω, όταν φτάνουν στα πώ δεν υποβάλλουν επίσημη αίτηση ασύλου. Το Δουβλίνο δεν ισχύει, δεν ισχύει τίποτα και η μόνη λύση θα ήταν να ήμασταν ευρηματικοί όπως ήταν και το ανώτατο δικαστήριο στη Μεγάλη Βρετανία σε μια σχετική υπόθεση όπου δυστυχώς όμως αυτά δεν ισχύουν και δεν έχει προστασία. Τώρα για την οικογενειακή επανένωση δεν πρέπει υποχρεωτικά ο μηχανισμός με κατάσταση να οδηγεί στην οικογενειακή επανένωση. Αλλά αυτό έχει γίνει τώρα προτεραιότητα λόγω του άρθρου 7 διάταξη, τέλο πάντων δεν ακριβώ, λέω μιλήτρια, αλλά τέλο πάντων έχουμε το δικαίωμα βάσει χάρτα για την, για την οικογενειακή ζωή. Και αυτό ακριβώς βεβαιώνει την κυριαρχία αυτού του άρθρου. Δηλαδή η επανένωση θα πρέπει να είναι προς το συμφέρον των παιδιών και αυτό τονίζει ακριβώς την αλλοεξάρτηση μεταξύ διαφόρων μελών της οικογένειας και την χρήση αυτών των οικογενειακών σχέσεων για τη διατήρηση οικογενειακής ενότητας. Οπότε θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος για να μειωθούν ακριβώς αυτές τις μεταφορές λόγω ε, Δουβλίνου όσον αφορά τις ε, επανενώσεις. Υπάρχει δηλαδή κάποιο υπογείμενο λόγο για την καθυστέρηση αυτή. Τώρα για τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησαμε για τη μελέτη, θα το αφήσω στην ΑΤΑΣ αυτό να το παρουσιάσει και θα επανέλθω στην παρακράτηση ατόμων στα hot spots στην Ελλάδα. Αυτό που συνέβη είναι ότι μετά την ε, σύναψη της συμφωνίας με την Τουρκία Είχαμε μια μεταρρύθμιση το 16 τον Απρίλιο στην ελληνική νομοθεσία ώστε να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα από τη συμφωνία με την Τουρκία επί τόπου. Οπότε όσοι κατέφταναν στα hot spots μετά την 20η Μαρτίου του 2016, ανεξάρτητα από το αν είχαν δικαίωμα κατάσταση δεν λάβαναν τη δυνατότητα αυτή να, να περιληφθούν σε αυτό το πρόγραμμα κατάσταση. Και πρέπει να πω ότι αυτό είναι παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, γιατί δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο ανεξαρτήτως ημερομηνία. Και αν παραμείνουμε στην τεκμηρίωση του δικαστηρίου, η συμφωνία με την Τουρκία δεν αφορά κάτι το οποίο προβλέπεται από τις συνθήκες, οπότε δεν θα πρέπει να επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας της συμφωνίας, η εφαρμογή της. Οπότε νομίζω ότι έχουμε ξεκάθαρα να κάνουμε μια παραβίαση τη κοινοτική νομοθεσία. Και το δικαστήριο του Στρασβούργου επίσης, αποφασίζοντας για τις συνθήκες υποδοχής ή τις ε, συνθήκες ασύλου, είπε ότι αυτό αποτρέπει ε, τον επαναπατρισμό Είχαμε μια υπόθεση στο δικαστήριο του Στρασβούργου για αυτό το θέμα. Δεν έχει σημασία λοιπόν αν ε, η Τουρκία αποτελεί παράδεισο για αυτούς τους ανθρώπους που είναι ευάλωτοι μια μεταφορά, μια μετακατάσταση υποχρεωτική με μέσα βίας θα πρέπει να αποφεύγεται. Και τέλος, για την υποχρέωση να υπογράψουν έντυπα που απαλλάσσουν ή αποτρέπουν τους δικαιούχους για δικαιώματα προσφυγής. Νομίζω ότι αυτό είναι μια αυθαιρεσία. Αν διαβάσετε ακριβώς ε, τον ορισμό ε, στο άρθρο 54 της Ταμείου κάρτα, Κάρτας των Αυθαιρεσιών, περί αυτού πρόκειται. Και τέλος, για τις επιδόσεις της Ιταλίας, η οποία έχει αναλάβει πολύ μεγάλο μερίδιο από, αυτό της, από, από αυτό που της αναλογεί και έχει λάβει πολύ σοβαρά την ρήτρα ελεγγύης ως νομικά δεσμευτική. Έκανε λοιπόν πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός από την Ελλάδα. Οπότε νομίζω ότι δεν θα πρέπει να πιέζουμε την Ιταλία και την Ελλάδα να συνεχίσουν να το κάνουν. Πάντως, για το σχόλιο μου σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου, δεν θεωρώ ότι είναι θετική. Νομίζω ότι αποτελεί μια επαναυποχώρηση όσον αφορά την προστασία των υποψηφίων προς άσυλο και των προσφύγων. Ένα ενδεχόμενο θετικό, αν διατηρηθεί αυτό το τμήμα της αντίστοιχης πρόσφατης, με πρόταση είναι ότι οι μετεκαταστάσεις θα είναι τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου Δηλαδή θα διατηρηθεί μια νοοτροπία, ένας τρόπος ε, σκέψης που θα θεωρεί ακριβώς την διαδικασία ασύλου ως κάτι το οποίο θα εκκινεί από αυτές τις συνθήκες. Αν λοιπόν υπάρχει κάτι θετικό, θα είναι από αυτή τη μεταρρύθμιση, θα είναι ότι ενσωματώνει την αρχή μετεγκατάσταση ω κάτι το οποίο θα θεωρείται φυσιολογικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συστήματο Ασύλου. Αλλιώ έχετε απόλυτα δίκιο. Το Δουβλίνο 4, αν εγκριθεί, θα δίνει προτερότητα στην προστασία σε σχέση με την συμφωνία με την Τουρκία. Αλλιώς η δεύτερη επιλογή θα είναι η προστασία στα hot spots. Οπότε και πάλι θα κάνουν την βαριά δουλειά η Ελλάδα και η Ιταλία. Οπότε κατά κάποιο τρόπο το βιβλίο σε αυτή την περίπτωση θα διονίζει τον θεσμό των ε, hot spots στην μεταβατική συμφωνία και η τελική προστασία κάπου αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν τελείως έκτακτη. σε σχέση με την διεθνή προστασία που παρέχει αυτή τη στιγμή η διεθνή ε, νομοθεσία, το οποίο είναι κάπω παράδοξο. Και Νατάσα. Για τη μεθοδολογία Έχω κάνει συνεντεύξεις ε, με εθνικά σημεία, ε, διεθνή σημεία επαφής ε, που με άτομα. Είναι μια έρευνα γραφείου. Και αυτό που προέκυψε είναι ότι τα κράτη-μέλη τα οποία μετεγκαθιστούν δεν μετεγκαθιστούν ανήλικους και άλλους ευάλωτους γιατί δεν έχουν τις εγκαταστάσεις για να το κάνουν. Φυσικά θα πρέπει να βασιστούν σε αυτά που τις λένε τα κράτη-μέλη. Ε, και αυτό που προτείνουμε λοιπόν στη μελέτη είναι να ελέγχε, ελέγχεται αν είναι πρόσχημα ή αν συμβαίνει όντως πραγματικά. Δηλαδή δεν υπάρχουν πραγματικές εγκαταστάσεις για να υποδεχθούν ε, τους ευάλωτους ετούντες άσυλο υπό το σύστημα με κατάσταση. Ή πω συμβαίνει κάτι άλλο επιπλέον πέρα από τις ε, έρευνε που κάναμε στην Ελλάδα και στην Ιταλία επιτόπου, κάναμε συντεύξει με τις αρχέ, τις φορείς και, τι τις ΜΚΟ ε, και να έρθουμε σε επαφή με τους ε, πρόσφυγες, αλλά δεν επισκεφτήκαμε κέντρο υποδοχή όμω. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε, γιατί οι μελέτε αυτές είναι θαυμάσίε, το ξέρω, και να μπούμε σε μεγαλύτερο βάθο, αλλά δυστυχώ έχουμε ακόμα ένα σημείο στη μέση διάταξη και είναι ένα σφάκελος που πρέπει και αυτόν να συζητήσουμε, γιατί είναι και εδώ η συγγήτρια. Σας ευχαριστώ για τη δουλειά σας, θα είναι πολύ χρήσιμη για το θέμα της μετεγκατάστασης και ελπίζω οι συνάδελφοι να χρησιμοποιήσουν αυτή τη θαυμάσια δουλειά του Policy Department. Φυσικά άκουσα τους επένους της κυρίας Σπινέλη, η οποία είναι ε, θαυμάστριά σας. Δεν υπάρχει ψηλότερος έπαινος από αυτόν. Ευχαριστούμε, Βιολέτα και φυσικά θα αναφερθούμε στη δουλειά σας στο μέλλον. Θα έρθει και η κυρία Σκάκελερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που κάθισαν μέχρι το τέλος της ημερησίας διάταξης και τώρα περνάμε σε, ένα, μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Ευχαριστώ τη Μάιτα Φάκο και την συνεισηγήτρια. Και τώρα θα εξετάσουμε ένα σχέδιο έκθεσης η ανακοίνωση της 5ης Ιουλίου και της, το πρόγραμμα της εργασίας του 2017 η Κομισιόν ε, είπε ότι θα αξιολογήσει το, το περιθώριο για ενωσιακή δράση για την προστασία των καταγγελόντων της λειτουργίας. Γι' αυτό κάνει μια μελέτη αντικτύπου αυτή τη στιγμή η Κομισιόν ε, και μια δημόσια διαβούλευση η οποία θα παρουσιαστεί στα τέλη του 2017 ούτως ώστε να συνεισφέρει ε, σε αυτό η Επιτροπή Γιούρη ε, κάνει μια έκθεση δίας πρωτοβουλίας για την προστασία των καταγγελόντων, όπου η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ετοιμάζει μια σημαντική γνωμοδότηση. Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ την εισαγωγή και θα δώσω το λόγο στη Μάιτο, Μάιτο η οποία περιμένει υπομονετικά και θα παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησής της. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αισθάνθηκα μεγάλη τιμή και ενδιαφέρον που άκουσα το προηγούμενο σημείο. Δυστυχώ δεν το άκουσα όλο. Ε, η έκθεση όμως που παρουσιάστηκε ήταν πολύ σημαντική, πολύ πολύ σημαντική. Και ήταν πολύ θετικό το ότι ήρθα εδώ και την άκουσα, όσο άκουσα. Τώρα, από πλευρά μου, αυτό που θέλω είναι να σας μιλήσω για την ανάγκη να εργαστούμε αμελητή πάνω σε αυτή την ε, γνωμοδότηση, για τη γνωμοδότηση. Για αυτούς που ε, είναι καθήλυνα αρμόδιοι στην Επιτροπή Γιούρη. Ε, από την περίοδο του Snowden, από τα Wikileaks, τα άτομα αυτά που μας βοηθάνε καταγγέλλοντας προβληματικές καταστάσεις, πλήττονται επειδή ακριβώς αποκαλύπτουν αυτές τις πληροφορίες ε, που ε, και πλήττονται, χάνουν συχνά την δουλειά τους, ε, πιέζονται, τα εκφοβίζουν, απειλές κτλ. δεν, έχουν ένα, δεν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που τους προστατεύει. Η ο διασυνοριακός χαρακτήρας κάποιων από αυτές τις, αυτά τα δικήματα, φοροδιαφυγή, διαφθορά, σημαίνει ότι και εμείς εμπλεκόμαστε και πρέπει κάτι να κάνουμε για αυτό το θέμα. Το Κοινοβούλιο ε, συμμετείχε και συζήτησε πολλές φορές ο, για την ανάγκη να κάνουμε κάτι για να προστατεύουμε αυτά τα άτομα, τα δικαιώματά τους, ε, κάποια σίγουρα κανάλια κτλ. Κάναμε επίσης μια ακρόαση στην Επιτροπή Πάνα και Γιούρη για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι εγώ γνωρίζω αρκετά άτομα τα οποία δεν προστατεύονται. Γιατί δεν προστατεύονται, γιατί μας βοήθησαν δίνοντας πληροφορίες για διάφορα πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Και έπρεπε να, παραδείγματο χάρη, ε, σε περίπτωση ενό ε, ενός ισπανικού αεροδρομίου για άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ένα άτομο ε, δούλεψε για τέσσερα χρόνια για να καταγγείλει τις καταστάσεις που πλήττουν, που παρεμποδίζουν τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα να κινηθούν. Ε, και η Κομισιόν, ε, η Κομισιόν εξετάζει αυτές τις παρατυπίες. Το άτομο αυτό που κατήγγειλε αυτά τα προβλήματα έχασε δουλειά του. Ε, αυτά, τα αυτά τα πράγματα έχουν μεγάλη αξία. Ε, καταγγέλουν παρατυπίες ε, για, ας πούμε, για περιπτώσεις κακομεταχείρισης επιβατών με προβλήματα, με αναπηρία κτλ. Είναι λοιπόν ευθύνη μας να βοηθήσουμε εκείνους που είναι καλοί πολίτες, που ξέρουν από, την αγωγή, αγωγή του πολίτη. Εμείς πρέπει να κάνουμε μία δουλειά μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας. Να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αστικές ελευθερίες. Η γνωμοδότηση που σας παρουσιάζω μιλάει και για την ε, εμπιστευτικότητα των, των στοιχείων αυτών, για την προστασία των δεδομένων. Ε, όλα αυτά αναφέρονται στην, στην Κάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αναμονήσουμε τα νομοθετικά πλαίσια για το θέμα αυτό και να ζητήσουμε από την Κομισιόν να θέσει ένα νομοθετικό πλαίσιο οριζόντιο, να δημιουργήσει νόμιμα ε, νομικά κανάλια για να διευκολύνει τη ροή των πληροφοριών ε, σε περίπτωση που υπάρχει ε, πρόβλημα στο δημόσιο συμφέρον και να υπάρχει πρόσβαση στο δικαίωμα της υπεράσπισης. Κάναμε μια αρχική ανταλλαγή απόψεων. Δεν είναι εύκολη η δουλειά αυτή. Έχουμε ασθενή νομική βάση. Θα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πρέπει να δουλέψουμε γρήγορα ούτω ώστε να μην έχουμε παρελκυστικές τάσεις, να μην παρατείνουμε το πρόβλημα αυτό. Πρέπει να το εξετάσουν οι συνομοθέτες. Και πρέπει να φτάσουμε σε μια οποιαδήποτε λύση με τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Είμαι πεπισμένη, παρόλα αυτά, ότι θα κάνουμε μια θαυμάσια δουλειά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Μαϊτέ. Το θέμα της νομικής βάσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε ένα σκιώδη μαζί μας, ο Ντένις. You're the S and D shadow. I'm so sorry, you are not listed on the... You are listed. Κύριε Κοστέλ, ε, ο κύριος Δεγιόν ήταν ε, σκιώδης των σοσιαλιστών. Συγγνώμη. Έχω κουραστεί, είναι πέμπτη. Παρακαλώ, ως σκιώδης των σοσιαλιστών, πείτε μας. Κύριε Κώστερ. Ευχαριστώ. Κανένα πρόβλημα. Μην ανησυχείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησης. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι ήρθε πια ο καιρός να προστατευτούν νομικά οι προφοριοδότες σε, ευρωπαϊκή, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και παρότι έχουμε ασκήσει μεγάλες πιέσεις στην Κομισιόν, η Κομισιόν δεν έχει ακόμη υποβάλει νομοθετική πρόταση. Είναι σκάνδαλο αυτό αν διώκονται, διώκονται δηλαδή οι πληροφοριοδότες, ενώ ταυτόχρονα οι μεγάλες εταιρείε επιδίδονται σε φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή, χωρίς καθόλου κυρώσεις. Ε, αυτό σημαίνει ότι κάτι είναι λάθος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. γιατί τους σοσιαλιστές είναι σαφές ότι οι πληροφοριοδότες, οι καταγγέλτες, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη παρατυπιών ή και παράνομων δραστηριοτήτων. Κατά τη γνώμη μας, οι καταγγέλτες είναι απαραίτητο στοιχείο για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της φοροδιαφυγής. Αποτελούν έναν πυλώνα απαραίτητο κατά τις διαφθορές και ε, ε, έναν τρόπο για να εξασφαλιστεί η λογοδοσία κυβερνήσεων και επιχειρήσεων. Και σε αυτές τις περιπτώσεις οι πληροφοριοδότες πολλές φορές αξιοποιούν ε, τον, ε, ε, μάλλον είναι ο, ο λόγος για τον οποίο αποκαλύπτονται πληροφορίες που κατά τα άλλα μένουν μυστικές. Γι' αυτό και οι πληροφοριοδότες είναι στοιχείο μιας εύρυθμης λειτουργίας της δημοκρατίας. Είναι στοιχείο της ελευθεροτυπίας, της ελευθερίας έκφρασης γνώμης για μια δημοκρατία. Γι' αυτό και πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εναρμονιστεί το επίπεδο προστασίας των πληροφοριοδοτών και αυτός, ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί με οριζόντια νομοθεσία. Όπω όπως και ο εισηγητής, είμαι και εγώ ε, υπέρ της δημιουργίας ενός συστήματος καταγγελιών και ενό συστήματος ευρωπαϊκού μηχανισμού προστασίας προκειμένου οι πληροφοριοδότες να μπορούν να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους. Τέλος θέλω να επισημάνω ότι οι πληροφοριοδότες ενεργούν με μεγάλο κίνδυνο και κόστος ε, προσωπικό, επαγγελματικό, οικονομικό, το οποίο πολλές φορές το επομίζονται μόνοι τους. Ας μην το ξεχνάμε αυτό και θα πρέπει επίσης να ε, εξετάσουμε και το, τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν. Τέλος, θέλω να προτείνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, απονέμει ένα βραβείο καταγγέλτη που θα μπορούσε να συμβάλλει ε, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης γύρω από τη σημασία που έχουν οι προφοροδότες στη δημοκρατία μας. Προσβλέπω στην καλή συνεργασία με την εισηγήτρια και ελπίζω να βρούμε μια ικανοποιητική λύση για, με απότερο στόχο την ε, αποτελεσματική προστασία των πληροφοριοδιωτών. Ευχαριστώ. Ενδιαφέρουσα αυτή η ιδέα ε, για το βραβείο. Ευχαριστούμε, Μάιτε. Ρομπέρτα θα μιλήσει εκ μέρου του ΕΛΚ και του Νίνο Μέλο. Ο Νούνο Μέλο θέλει να ζητήσει συγγνώμη για την απουσία του από τη σημερινή συζήτηση, ωστόσο ε, βρίσκεται σε επίσκεψη στην Πορτογαλία στο πλαίσιο της Επιτροπής ΠΑΝΑ. Θα ήθελα παρόλα αυτά να ευχαριστήσει την εισηγήτρια για την γνωμοδότησή της και για την στάση της, την επικοδομητική της στάση προκειμένου να εξευρεθεί συμβιβασμό. Πέραν τη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών και την ανάγκη ενισχυμένης συνεργασία, ο Σκιώδη μα πιστεύει ότι ένα από τα εργαλεία για την καταπολέμηση τη διαφθορά και του οργανωμένου εγκλήματο είναι ακριβώ η ύπαρξη των πληροφοριοδοτών. Το να ενθαρρύνονται λοιπόν οι εργαζόμενοι να καταγγέλουν παρατυπίες και να προστατεύονται όταν το κάνουν είναι τρόπος ε, για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος στον δημόσιο τομέα, οι πληροφοριοδότες μπορούν να βοηθήσουν στην αποκάλυψη κατάχρησης δημόσιου χρήματος, διαφθοράς και άλλων διασυνοριακών εγκλημάτων που στρέφονται κατά των εθνικών και ενωσιακών συμφερόντων. Είναι σημαντικό οι μυστικές πληροφορίε να μπορούν να αποκαλύπτονται και γι' αυτό είναι σωστό να μπορεί κανεί να αποκαλύπτει κακομεταχείριση, κακοδιαχείριση και παρατυπίε. Ε, τα πρόσφατα σκάνδαλα ε, αποκαλύφθηκαν ακριβώς χάρη στους ε, πληροφοριοδότες, όπως αποδεικνύουν και τα έγγραφα του Παναμά, τα οποία χάρη στους πληροφοριοδότες επέτρεψαν τη διενέργεια ευρύτερων δημοσιογραφικών ερευνών. Ο κύριος Νέλο είναι στη διάθεση της εισηγήτριας και όλων των άλλων σκληροδών για μια επικοδομητική συνεργασία. Ευχαριστώ και για την εκπροσώπηση του σκιώδους Ντένις ε, Ντεγιόν για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στην συγκίτρια. Καταρχάς, πολύ καλή η σύνταξη ευφυής και πολύ χρήσιμη. Τα σχόλια μου αφορούν δύο μέρη. Ένα γενικό επειδή και εγώ είμαι εισηγητής για παρόμοιο θέμα και αυτή τη βδομάδα είχαμε κάποιες ενδιαφέρουσες συνεδριάσεις. Η Επιτροπή είπε ότι θα υποβάλει τις απόψεις, απόψεις της το Σεπτέμβρη μετά τα ευρήματα οπότε μπορούμε να συσχετίσουμε αυτή την γνωμοδότηση με αυτή τη διαδικασία ώστε να δώσουμε ένα κίνητρο στην Κομισιόν ώστε να το θεωρήσει υψηλότερης προτεραιότητας. Μετά, είχα μια έκθεση της Επιτροπής Ολόκληρου του που εγκρίθηκε τον Φλεβάρη και είχαμε και ψήφισμα σε σχέση με την προστασία αυτών των ανθρώπων όταν δίνουν πληροφορίες για οικονομικά συμφέροντα. Νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο θα ήταν ενδιαφέρον ή χρήσιμο στο ψήφισμα να αναφερθούμε άμεσα ή έμεσα ας πούμε στον ορισμό του πληροφοριοδότη. Ε, εμείς έχουμε θετήσει ένα έγγραφο που μιλάει για πληροφορίε που είναι 100% αληθείς αλλά και ότι αυτός ο πληροφοριοδότης θεωρεί ότι είναι αληθείς αυτές τις πληροφορίες ώστε να μην διώκονται σε περίπτωση που οι πληροφορίες δεν είναι αληθείς αλλά αυτοί είχαν καλή πρόθεση αρχικά. Βλέπω επίσης ότι στο ψήφισμα είπαμε χρειαζόμαστε κάποιες ανεξάρτητες αρχές και χθεσινές πληροφορίες από την διαμεσολαβήτρια λένε ότι προτίθεται να το εξετάσει αυτό. Δηλαδή ένας τρόπος διευκόλυνσης των πληροφοριωτών είναι το να έχουν κάποιο ρόλο που να σχετίζεται με, τον διαμεσολαβητή. Αυτό, γι' αυτό είναι ανοιχτό ο διαμεσολαβητής και πρέπει να το διερευνήσουμε. Επίσης, νομίζω θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι πληροφοριοδότες δεν μπορούν να είναι προσωπικό κάποιων ευρωπαϊκών θεσμών. Χρειάζεται προστασία. Γιατί βλέπουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις λείπει. Οπότε πρέπει να υιοθετήσουμε κάποια μέτρα που θα ήταν καλό να υιοθετηθούν νομικά. Δεν ξέρω πώς, ίσως να μην είναι εδώ το κατάλληλο μέρος, αλλά μας απογοήτευσε το αποτέλεσμα της οδηγίας για τα εμπορικά μυστικά. Επειδή εκεί ακριβώς είδαμε ότι δεν υπάρχει προστασία 100% για αυτά τα άτομα και αυτά ακριβώς χρειαζόμαστε κάτι εδώ. Να υπάρχει δηλαδή ένα είδο διπλωματικού κειμένου που να παραπέμπει σε αυτό, χωρί βέβαια να το μετατρέψει σε κάτι πολύ επίμαχο. Ευχαριστώ. Το ECDR. Μήπω κάποιο άλλο θέλει το λόγο. Κατερίνα, θες ε, δύο λογάκια η Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ, πολύ σύντομα, γιατί και εγώ εργάστηκα σε άλλη για αυτό το θέμα και γνωρίζω την Ιταλική εμπειρία και τη σημασία που έχουν οι συνεργάτες οι οποίοι μπορούν να παράσχουν σημαντικές ε, πληροφορίες σε σχέση με μεγάλα δικήματα ότι ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με απάτες, μορφές διαφθοράς, οικονομικά συμφέροντα, εγκλήματα δηλαδή οικονομικής φύσεως πολύ σημαντικά. Οπότε συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι και του συγχαίρω για τη δουλειά που έχει γίνει, αλλά κυρίως για τη δουλειά που θα κάνουν. Είναι σημαντικό να υπάρχουν άτομα τα οποία από μέσα θα μπορούν να δίνουν πληροφορίε, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτών των εγκλημάτων. Βεβαίως θα πρέπει να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι σημαντικό επίσης να έχουμε και ένα κοινό ορισμό αυτών των πληροφοριοδοτών πανευρωπαϊκά ώστε να αναρμονιστούν και οι νομοθεσίες. Και είναι σημαντικό βέβαια να τους δίδεται η προστασία την οποία αναφέραμε, ώστε να αποφεύγονται οι εκβιασμοί και οι αρνητικές επιπτώσεις στην σταδιοδρομία τους ή στην καθημερινότητά τους. Είναι σημαντικό αυτό και για ένα άλλο λόγο νομίζω. Επειδή θα πρέπει οι πολίτες να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους στα θεσμικά όργανα. Ιδιαίτερα αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και εργάζονται σε αυτού του τομεί. Οπότε συμμερίζομαι αυτά που υπόθηκαν και είναι ε, σημαντικό, όπω είπε η συγγήτρια, να επιταχύνουμε τη διαδικασία για αυτό το θέμα, γιατί θα αποτελέσει πραγματικά ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των οικονομικών εγκλημάτων. Αυτό ήθελα εγώ να πω και να τονίσω ότι συμμερίζομαι απόλυτα τη δουλειά που γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Κατρίν. Ναι, θέλετε να ολοκληρώσετε. Ναι, σας ευχαριστώ όλους τα συγκήτρια για την ευαισθησία και την ε, βούλησή σας για συνεργασία αλλά και για τα σχόλιά σας. Και να σας υπενθυμίσω ότι στις 23 του ήλιου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες, οπότε καταθέστε Ελπίζω να πάμε γρήγορα και να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα και ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Τι ωραίο να έχουμε τέτοιε ωραίες συζητήσει για το τέλος. Ευχαριστώ συνάδελφοι, ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ και το προσωπικό και καλώς το Κυριακό. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τίποτα στα διάφορα? Όχι. 26 Ιούνιου που επόμενη συνάντησή Ευχαριστώ συνάδελφοι. Γεια σα.